Όπως βλέπετε, καλημέρα σας βέβαια, δεν είμαι η Καρίμα Νταλή, αλλά θα προεδρεύσω σήμερα την Επιτροπή των Μεταφορών. Και καλά, μη φοβάστε, μη φοβάστε. Βλέπω να φοράτε ακουστικά γιατί θα τα πω στα αγγλικά. Συνάδελφοι, πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης και θα συζητήσουμε τα της μελέτης ε, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε το τοπίο που ισχύει τώρα, να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες για τον κλάδο στην Ευρώπη. Καλωσορίσατε ορίσατε κύριε Τσερπίτσκης και κυρία Φατσίνο στην Επιτροπή μας. Να δώσουμε πρώτα το λόγο σε εσάς για πέντε λεπτά στον καθένα και κατόπιν να συζητήσουμε. Να λάβουν το λόγο πρώτα οι συντονιστέ και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κυρία Φατσίνο, εσεί έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτέ, είναι τιμή μα που σήμερα είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε αυτήν την ε, μελέτη για τις ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφος και εγώ ερχόμαστε από το Ίδρυμα Copenhagen Economics και παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες συμβουλών και άλλες. Έχουμε τρεις άξονες να σας παρουσιάσουμε το θέμα μας. Πρώτα-πρώτα τις εξελίξεις, κατόπιν τα προβλήματα, προκλήσεις, ευκαιρίες, ε, την ανταπόκριση από την πολιτική και τέλος τις προτάσεις μας. Πρώτα-πρώτα να σας πούμε πώς έχει το πλαίσιο για ε, το ρυθμιστικό περιβάλλον. Πρώτα-πρώτα, έχουμε από το 1997 ε, την ε, οδηγία για την εναρμόνιση της ενίας αγοράς, για τη βελτίωση επίσης των υπηρεσιών. Ε, επίσης, για το πώς θα ανοιχτεί στον ανταγωνισμό ο κλάδος, έχει τροποποιηθεί δύο φορές αυτή η οδηγία. Τελευταία φορά το 8. Και τώρα ξεκινούμε ένα νέο νομοθετικό κύκλο για περαιτέρω τροποποίηση από την Κομισιόν. Το 2018 είχαμε τον κανονισμό για τις διασυνορικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Αυτός ο κλάδος που συζητούμε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχει τζίρο 80 δις, περισσότερο από το ΑΕΠ Λιθουανίας και Λετωνίας απασχολεί 7 εκατομμύρια, ε, περισσότερους δηλαδή από τους κατοίκους της ε, Κροατίας και έχει ανάπτυξη 2,4% κάθε χρόνο, δηλαδή περισσότερο τον πληθωρισμό. Υπάρχουν πολλές αλλαγές όμως που προέρχονται από τη ψηφιακή τεχνολογία. Πρώτα-πρώτα ο κόσμος και οι εταιρείε επικοινωνούν περισσότερο ψηφιακά, όλο ένα και περισσότερο και βλέπουμε οι επιστολές συνεχώς να μειώνονται από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι περισσότεροι ψωνίζουν ε, από το ίντερνετ, οπότε βλέπουμε να αυξάνονται τα δέματα που παραδίδονται. Βλέπουμε επομένως εξέλιξη του ανταγωνισμού, ε, έχουμε τους ε, βασικούς παρόχους στα κρατή-μέλη, που είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν ανταγωνιστές ψηφιακοί και ό,τι παλιά γινόταν ε, με επιστολές, τώρα γίνεται με το email, ε, με το ίντερνετ. Και βλέπουμε ότι είναι λιγότεροι τώρα οι πάροχοι από τους ε, παρόχους του ίντερνετ. Και η συνέπεια είναι ότι οι επιδόσεις αυτών των υπαρχόντων παρόχων συνεχώς μειώνονται. Τέλος, έχει περισσότερο ο κόσμος τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι αλλαγές ε, στο μείγμα προϊόντων ε, σημαίνει ότι έχουμε όλο ένα και λιγότερες επιστολές, καλύτερο για το περιβάλλον, ε, γιατί ένα δέμα είναι 12 φορές περισσότερο διοξίδιο από μια επιστολή και θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι αληθείς επιπτώσεις. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να παραδίδεται στον καταναλωτή ε, το δέμα παρά να πάει να το ψάξει, να το πάρει ο καταναλωτής. Και τώρα για τις ε, προκλήσεις και τις ευκαιρίες έχει τη ο συνάδελφος. Είναι τιμή μου κύριοι βουλευτές να σας παρουσιάσω τη μελέτη μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε στη μελέτη μας ότι αυτός ο κλάδος έχει πάρα πολλές προκλήσεις, προβλήματα να αντιμετωπίσει. Βασικά πρόκειται για τη μείωση των επιστολών και ε, αυτό που τελεί μια απειλή για τις καθολικές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι θέμα μόνο τα χρηματοοικονομικά ορισμένων εταιριών. Το θέμα είναι το ότι έχουμε κάποιους ευάλωτους χρήστες που εξαρτώνται από αυτές τις υπηρεσίες και είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον ε, κλάδο. Οπότε είναι περίπλοκη η κατάσταση αυτό γιατί δεν είναι μόνο θέμα το νομοθετικό περιβάλλον ε, είναι και άλλα ζητήματα όπως οι πολιτικές για το περιβάλλον, όπως η νομοθεσία για τον ΦΠΑ, οπότε και στην ε, μελέτη μας προσπαθούμε αυτά να τα δούμε όπως είναι αλληλένδετα. Επίσης υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για τον κλάδο. Αυξάνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και αυτό είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τους παρέχους για να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας και όμως διαπιστώσαμε ότι μόνο πολύ λίγοι από τους παρόχους τα κατάφεραν να αντικαταστήσουν τη μείωση των επιστολών ε, με την αύξηση των δεμάτων. Και αυτό βασικά γιατί είναι πολύ άγριος ο ανταγωνισμός όσον αφορά τα δέματα. Άλλη ευκαιρία είναι το δίκτυο και το brand value το οποίο έχει σχέση με αυτό το ζήτημα και αυτό αφορά κάποιες χώρες που είναι καλύτερες από άλλες σε αυτό, Φερρυπίν. Το Μπιπόστ και το γαλλικό ταχυδρομείο τα πάνε πολύ καλά σε Βέλγιο και Γαλλία για αυτές τις υπηρεσίες και επίσης διαπιστώσαμε αυξανόμενο ενδιαφέρον από άλλες χώρες για να διδαχθούν από τις καλές αυτές πρακτικές εκείνων των χωρών. Επίσης, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, αυτές μπορούν να φέρουν περισσότερη αποτελεσματικότητα και νέες υπηρεσίες στην αγορά. Αυτές οι τρεις ευκαιρίες διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου. Οπότε και είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι θα έχουν την ικανότητα και την ευελιξία να τις αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Όντως, αν ρίξει κανείς μια ματιά τι γίνεται στις διάφορες χώρες, τι προβληματικές υπάρχουν. Η λέξη κλειδί είναι η ευελιξία σε κάποιες χώρες, γίνεται κουβέντα για το πόση ε, ελευθερία θα πρέπει να έχουν οι πάροχοι για την προσαρμογή των υπηρεσιών, του δικτύου τους, στις αλλαγές όσον αφορά την ζήτηση και σας υπενθυμίζω ότι η σχετική οδηγία έχει κάποιες μήνυμου προϋποθέσεις για τα κράτη-μέλη. Φερρυπίν, πόσο συχνά θα πρέπει να πηγαίνει στα σπίτια κάθε εβδομάδα ο ταχυδρόμος και λέει η οδηγία πέντε μέρες τη εβδομάδα. Αλλά σε κάποιες χώρες υπάρχει νομοθεσία που επιβάλλει έξι μέρες τη βδομάδα, δηλαδή παραπάνω από την όρμα. Οπότε συζητάμε για τις ελάχιστε προποθέσει που είπαμε ότι είναι αυτές. Πέντε μέρες και άρα, να, τι συζήτηση υπάρχει για το θέμα επίσης. Ευελιξία στην τιμολόγηση. Επίσης διαμορφώνεται μία τάση να εξετάζεται η βιωσιμότητα των υπηρεσιών αυτών και να έχει προτεραιότητα έναντι άλλων στόχων όπως την βελτίωση του ανταγωνισμού. Και έρχομαστε τώρα στο τελευταίο μας σημείο της συστάσης μας. Η βασική μας πρόταση προς εσάς είναι να λάβετε υπόψη ότι τα κρατημέλη έχουν διαφορετικές ανάγκες, διότι έχει το καθένα διαφορετικά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Ιστορικά υπήρχε μονοπόλιο στην αγορά και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το μονοπόλιο γιατί αν συνεχίζει αυτό να ισχύει σε κάποιες χώρες οι οικονομολόγοι λέμε ότι οποιαδήποτε επανέμβαση στην αγορά θα πρέπει να εστιάζεται σε κάποιο είδους σαφές καθορισμένο πρόβλημα της αγοράς. Και σε κάποιες χώρες το βασικό πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα των καθολικών υπηρεσιών. Οπότε για αυτές τις χώρες το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να δίνει αρκετή ευελιξία για την, για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Τέλος, αυτό το οποίο τελευταία διαπιστώνουμε είναι ότι η ευελιξία δεν αρκεί ούτω ώστε να υπάρχει βιώσιμη παροχή αυτών των υπηρεσιών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις χώρες η κρατική νομοθεσία να εγγυάται όλα αυτά, δηλαδή τις παροχές των υπηρεσιών αυτών εις τους πιο ευάλωτους ε, χρήστες. Εδώ ολοκληρώνει την παρουσίασή μας και είμαστε έτοιμοι για τις ερωτήσεις σας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Χατσίνο και, και κύριε Τσεπίκης. Θα έχουμε τώρα τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων του συντονιστές θα δώσω τον λόγο. Ο κύριος Μαρινέσκου δεν είναι εδώ. Ο κύριος Φάμπρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας. Η μελέτη αυτή μου θυμίζει τα νιάτα μου. Ήμουν ε, εισηγητής, ε, εισηγητής στην πρώτη ταχυδρομική οδηγία και στη δεύτερη και τρίτη, οπότε έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Τότε το σκεπτικό μας ήταν... Δεν ξέρω αν διάβασα καλά τη μελέτη. Ναι, η πρόθεσή μας ήταν οπωσδήποτε να επιτύχουμε κάτι το οποίο δεν ε, επιτύχαμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα έχουμε ε, πιο απομονωμένες εθνικές αγορές από ό,τι είχαμε τότε. Και βεβαίως αυτό έπαιξε ρόλο κάτι το οποίο αναφέρατε στην μελέτη σας, δηλαδή ότι υπήρχαν κράτη-μέλη που χρησιμοποίησαν τις ε, δυνατότητες της παγκόσμιας ταχυδρομικής σύμβασης για να εμποδίσουν τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς κάτι το οποίο σημαίνει ότι σήμερα έχουμε τιμές για διασυνοριακά που είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν από την πρώτη οδηγία. Οπότε το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε για να καταλήξουμε σε μια εσωτερική αγορά και να μην έχουμε 28 ή 27 προσεχώς εθνικές ε, ταχυδρομικές αγορές. Δεύτερον, μιλήστε για την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Αν το δούμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πολύ περιορισμένες ε, πέντε μέρες και κάποιες ποιότητες, κάποιες υποχρεώσεις ποιότητας. Όλα τα άλλα είναι εθνικές υποχρεώσεις στη χώρα μου ας πούμε. Το θέμα ρυθμίζεται πάρα πολύ πόσο πρέπει να απέχει ένα ταχυδρομικό κουτί από τον τελευταίο κάτοικο που είναι δύο χιλιόμετρα ας πούμε. Βεβαίω αυτό σημαίνει μεγάλο κόστος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο όρισε ο Ευρωπαίος νομοθέτης. Ε, βεβαίως ε, σημαίνει ότι μεταφέρθηκαν αυτές οι υπηρεσίες στο ταχυδρομείο. Οπότε διατηρήθηκε το μονοπόλιο γιατί το κράτος ε, αναθέτει στα ταχυδρομεία κάποιες ε, υπηρεσίες. Παλιότερα μετέφεραν και τις συντάξεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δραστηριότητες που δεν κάνει το κράτος αλλά γίνονται στο ταχυδρομείο και έτσι γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα ε, για τους ανταγωνιστές. Αυτό όμως ε, δεν έχει σχέση με την ευρωπαϊκή ε, υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Λοιπόν, θα πρέπει το ταχυδρομείο πράγμα να επικεντρωθεί σε αυτό το οποίο είναι, δηλαδή ταχυδρομικές υπηρεσίες και μετά ε, υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρατε. Το είδαμε ήδη στην πρώτη οδηγία και στην πράσινη βίβλο τέλη δεκαετίας του 80 ότι είχε απελευθερωθεί σε μεγάλο βαθμό ο τομέας των πακέτων και παραμένει βεβαίως ε, απελευθερωμένος. Υπάρχει ένα ζήτημα βεβαίως όσον αφορά τις διεθνείς αποστολές πακέτων Λοιπόν, το ότι αναπτύσσεται ο τομέας των δεμάτων είναι θετικό ή αρνητικό παράδειγμα. Αναφερθήκατε επίσης στο θέμα της ε, ε, επιδότησης, ε, σταυροειδούς επιδότησης. Ειδικά σε σχέση με τις διατάξεις που γράψαμε στην τρίτη οδηγία έτσι ώστε τα κέρδη του μονοπωλίου να μην μεταφέρονται αυτομάτως στον ανταγωνιστικό τομέα των ταχυδρομείων. Α, γιατί τελικά τι θα πρέπει να κάνουμε, να επανέλθουμε στο παλιό μονοπόλιο ή τη δική μου την άποψη να έχουμε μια εσωτερική αγορά στις ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Φερμπέρ, για το μικρό, τη μικρή ιστορική αναδρομή που μας κάνατε. Ο κύριος Ντάνιλσον για τους σοσιαλιστές και μετά το Ινιού. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ για την ωραία παρουσίαση. Τονίσατε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα εστιάσω σε κάποια διαφορετικά που υπάρχουν στη δική μας έκθεση, αλλά όχι τόσο πολύ στην παρουσίασή σας. Γιατί με την ψηφιοποίηση και το αυξανόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχει ε, αυξημένη ζήτηση για παράδοση πακέτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, όπως είπατε, υπάρχει και αυξημένος ανταγωνισμός στον τομέα. Αυτός ο ανταγωνισμός συχνά είναι προς του καταναλωτή, αλλά μερικές φορές είναι και εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Σε διάφορες ε, χώρες, όπως την ε, δική μου ας τη χώρα, που έχουμε κρατικές ε, υπηρεσίες, καθολικής, καθολικές υπηρεσίες, χρησιμοποιούνται άλλοι άλλε εταιρείε για την παράδοση, μη κρατικέ, για την παράδοση των πακέτων. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα με του εργαζόμενου. Ε, πολύ ωραία, αυξημένο ανταγωνισμό, και... αλλά δεν θα πρέπει να είναι, πολλές, πολύ συχνά είναι η προσόφλωση του καταναλωτή, δεν θα πρέπει να είναι ει βάρο των ε, εργαζομένων. Έχουμε διάφορες συμβάσεις εργασίας σε αυτές τις περιπτώσεις, ε, διάφορα μοντέλα εργασίας. Πώς τα ρυθμίσουμε αυτά, τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα εμείς ως πολιτικοί για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τέτοιες διαφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης ε, πιο ευρέως τι άλλο χρειάζεται. Κάνατε κάποιες συστάσεις, αλλά ποιε είναι οι συγκεκριμένες ε, συστάσεις προς τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς τους πολιτικούς. Ευχαριστώ κύριε Ντάνιλσον. Από το Ρινιού. Θα μιλήσω εγώ, σύντομα. Είμαι Γερμανός. Την κάναμε σε κάποιες ε, περιοχές υπαίθρα τη συζήτηση. Συχνά οι ταχυδρομικέ υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζονται κάθε μέρα. Αλλά ο κόσμος ε, διερωτάται αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μερικές φορές διερωτώ με. Αν ε, με το μονοπόλιο θα είχαμε πιο... θα λειτουργούσε καλύτερα το πράγμα. Ας πούμε, οι περιοχές της υπαίθρου στην ε, Γερμανία είναι μια ειδική κατηγορία. Ίσως δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ε, σε άλλες χώρες τι συμβαίνει. Έχουμε παράδοση και εξασφάλιση υπηρεσιών στις ε, περιοχές της υπαίθρου 5 ή 6 μέρες τη βδομάδα. Και τι θα συμβεί κάτι γνώμη σας αν καταστρέψουμε τα μονοπόλια, ε, θα έρχονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στις περιοχές υπαίθρου κάθε μέρα. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συντάχτες για την καλή τους έκθεση. Δείχνει ότι το ταχυδρομείο παράγει, παραδίδει διάφορες υπηρεσίες. Όχι μόνο παραδίδει, είναι και κοινωνικέ υπηρεσίε, ειδικά για του ηλικιωμένου στην Ήπεθρο. Ξέρουμε ότι το ταχυδρομείο είναι ο σύνδεσμό του με το κράτο. Ο κόσμο το θέλει το ταχυδρομείο, θέλει να συνεχίσει να υπάρχει. Επίση, μιλήσατε για την περιβαλλοντική διάσταση και επίπτωση των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σε δραστηριότητες λιανεμπορίου που γίνονται πια επιγραμμικά. Και ο κίνδυνος να αυξηθεί το αποτύπωμα ε, του άνθρακα, εάν ένα μικρό πραγματάκι, ας πούμε, παραδίδεται σαν τεράστιο κουτί. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποιες συνέργειες. Ε, πέρα έξω από τις πόλεις και τις μεγάλες πόλεις, το κράτος έχει διάφορες μεταφορικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες για τα πακέτα και ε, τα γράμματα, ε, χάρη μεταφορές ε, στα σχολεία, ε, υπηρεσίες ε, μεταφοράς ε, ασθενών στα νοσοκομεία κτλ. Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε κάποιε συνέργειε ανάμεσα αυτά τα επίπεδα. Σε ορισμένε ε, χώρε έχουμε το ταχυδρομικό λεωφορείο που εξασφαλίζει και την παράδοση του ταχυδρομείου, αλλά μεταφέρει και κόσμο. Έτσι έχουμε εξοικονόμηση προς όφελος του περιβάλλοντος. Αλλά επίσης βοηθάμε και τις απομακρυσμένες περιοχές υπαίθρου, ας πούμε, που πλήττονται από τη μείωση των κρατικών υπηρεσιών. Ίσως θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και συμπερασματικά σας ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ε, περνούν από μια περίοδο ταχαίων αλλαγών και για να επιβιώσουν θα πρέπει να καινοτομήσουν. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή την καινοτομία, ούτω ώστε το κράτος να μπορεί να παράσχει αυτές τις πολύτιμες υπηρεσίες. Ευχαριστώ κύριε Καφ. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Λεσάντε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Να υπενθυμίσω τη σημασία του ταχυδρομικού τομέα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το οικονομικό βάρος του κλάδου και δεύτερον, την αποστολή του για τις καθολικές υπηρεσίες που καθορίζεται από μια ευρωπαϊκή οδηγία. Θέλουμε ποιοτικέ ε, ταχυδρομικέ υπηρεσίε σε μόνιμη βάση σε κάθε σημείο της επικράτειας, σε προσιτέ τιμέ για όλου τους χρήστε. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό βάρο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κλάδου, οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε είναι 79 δισεκατομμύρια ευρώ και ε, δίνουν δουλειά σε 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ο τρίτος εργοδότης στη χώρα. Είναι το πρώτο εμπορικό δίκτυο. Έχουν το πρώτο εμπορικό δίκτυο. Καταλαβαίνουμε χάρη σε αυτά τα νούμερα την ε, σημασία και, το, και την πίεση που του ασκούν ορισμένες αμερικάνικες εταιρείε. Ε, είναι μια κερδοφόρα αγορά που θέλουν να ανοίξουν περισσότερο στην, ε, στον ανταγωνισμό. Ξέρουμε όμως ότι το ταχυδρομείο εξασφαλίζει τις καθολικές υπηρεσίες ούτω ώστε να καλύψει ανάγκες του κόσμου δίνει και μοιράζει παντού ε, πακέτα και επιστολές. Ε, επίσης, ε, παράσχει ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλους. Εξασφαλίζει αυτή την παρουσία του κράτους και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και μειώνει τις ανισότητες ανάμεσα στις αστικές και περιοχές και στις υπόλοιπες. Θα ήθελα λοιπόν να δείξουμε μεγάλη προσοχή γιατί αυτές οι λειτουργίες και αυτή η αποστολή είναι εκ των όνων κάνευ. Συμφωνούμε όλοι επ' αυτού. Ε, αλλά συχνά δεν είναι κερδοφόρε αυτές οι υπηρεσίες που παρέχει το αχυδρομείο και σε καμία περίπτωση ο ιδιωτικό κλάδο θα αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες. ECR. Ε ο κύριος Ζουσό θέλει το λόγο. No. Uh, Κυρία Ντάλη, για την ΚΟΕ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ανθρώπους που έκαναν την μελέτη που παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταχυδρομείων. Και στην Ιρλανδία επίσης από όταν άνοιξε ο κλάδος. Είχαμε τεράστιες μετακινήσεις ε, και διαδηλώσεις από πλευράς μας για να προστατεύσουμε τα ταχυδρομεία μας ε, που αποτελούν ε, σημείο αναφοράς ε, στις αγροτικές κοινότητες μοιράζουν και τις συντάξεις και είναι νομίζω ανεκτήμητες αλλά αν δούμε στην Ευρώπη η μείωση του κόστους ε, των παρόχων της καθολικής υπηρεσίας και οδηγεί σε μείωση της απασχόλησης ε, εναλλακτική απασχόληση με χειρότερες συνθήκες εργασίας και χαμηλότερους μισθούς και βεβαίω υπάρχει η πρόκληση των ε, αντιπάλων χαμηλό κόστου. Το αναφέρατε και είπατε ότι πρέπει να το προσέξουμε αλλά όχι αρκετά. Δεν το τονίσατε αρκετά. Συνολικά θεωρώ ότι είχαμε αρνητικέ συνέπειε για τους εργαζόμενους των ε, παραδοσιακών ταχυδρομείων που έχουν υπονομευθεί από τους ε, ανταγωνιστές τους οι οποίοι χρησιμοποιούν ε, διάφορες ελαστικές μορφές εργασίας και να αναρωτιέμαι στο πλαίσιο αυτό ε, για το κατά πόσο θα πρέπει να υπερασπίσουμε τον κλάδο. Γιατί η περαιτέρω απελευθέρωση θα κάνει την κατάσταση χειρότερη. Βεβαίω ε, υπάρχει οδηγία, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τον κοινωνικό αντίκτυπο, κατά το οποίο δεν αναφέρουμε αρκετά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε σε έναν αγώνα και έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ενδιαφέρονται αυτά τα οποία είπατε και για το περιβάλλον. Αλλά ενδιαφέρον θα είναι το πώς ε, βλέπετε και αυτόν τον παραγόντα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Μινιός θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστούμε για ε, την παρουσίασή σας και συγχαρητήρια για τη μελέτη σας. Και χαίρομαι διότι ε, αυτή η μελέτη έλαβε υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των ε, εφαρμοστέων πολιτικών και επίσης να δούμε το θέμα της βιωσιμότητας του κλάδου και χρειάζεται η ευελιξία που αναφέρατε γιατί θα πρέπει αυτός ο κλάδος να λάβει υπόψη τις ανάγκες των πιο ευάλωτων χρηστών, δηλαδή αυτούς που μένουν στην Ήπεθρο και τους πιο ηλικιωμένους. Γι' αυτό σας λέω ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες σε κάποια χωριά όπως αυτό που προέρχομαι εγώ συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου και αυτών των ε, τοποθεσιών και επίση σε κάποιες ε, ζώνες όπου είναι αεροκατοικημένες εκεί αυτές οι υπηρεσίες ε, δεν είναι μόνο ότι δίνουν την ελογραφία, αλλά έτσι δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να αγοράζει εισιτήρια τρένου, ε, ή ε, έτσι μπορεί να πουλήσει ο κόσμος κάποια τοπικά ε, προϊόντα και όλα αυτά γίνονται με τις τεχνολογικές υπηρεσίες στην Ήπεθρο. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι προσπάθειες να αναγνωριστούν. Ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όταν φύγονται αυτές οι υπηρεσίες και να λάβουμε υπόψη, ε, μια που το συζητούμε και θα το συζητήσουμε εδώ, το θέμα των ε, δεμάτων που παραδίδονται με τα φορτηγάκια. Είναι το θέμα της αμεσότητος. Αυτό θέλει ο χρήστης από αυτό τον κλάδο. Και έτσι επομένως έχουμε και πιο σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον μια που όλοι έχουμε υποσχεθεί να συμβάλλουμε για την ε, πιο οικολογική μετάβαση, θα πρέπει να δούμε το πόσο κλάδος θα διακρίνεται από μια βιώσιμη κινητικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κριστιαμινιός. Τώρα, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Ποιος ε, θέλει τον λόγο πρώτος. Κύριε Τσαπίκης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις ε, μαζί. Υπάρχει σαφής ανησυχία για τις υπηρεσίες ε, κοινού συμφέροντος. Και βεβαίω ε, είναι σημαντικό ο αντίκτυπο του ανταγωνισμού. Υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να προλάβουμε τον αντικό αντίκτυπο. Ε, είναι σαφώς μια ενισχύ αλλά από την άλλη είναι και μια ευκαιρία για να βελτιωθεί η χρήση του δικτύου. Αυτό είναι το βασικό θέμα. <clears throat> Γιατί το μοναδιαίο κόστος ανεβαίνει και ανεβαίνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Ενώ οι τιμές δεν μπορούν να αυξηθούν ε, εξίσου γρήγορα, αφενός γιατί δεν θα είναι πρόσιτες. Και εφετέρου υπάρχει και ο παράγων ψηφιακών ε, υπηρεσιών. Αυτές είναι οι προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζουν τα ταχυδρομεία. Επίσης, Υπάρχουν ε, οι σκέψεις είτε για περαιτέρω ρύθμιση είτε για ε, απορρίθμιση. Και αυτό σχετίζεται με τους στόχους της πολιτικής. Και πρέπει να σκεφτούμε και πάλι ποιος είναι ο στόχος της ρύθμισης ούτως ή άλλως. Από την οικονομική σκοπιά είναι μια δύσκολη ερώτηση. Αλλά οπωσδήποτε μας δείχνει πώς λειτουργεί η αγορά, γιατί αν δούμε τις περιοχές της Υπέθρου, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ανταγωνισμό ακόμα ε, για τις υπηρεσίες ε, τις επιστολικές παρά το ότι ε, μπορούν οι εταιρείε να μπουν, είναι ελεύθερες. Αλλά δεν συμφέρει, δεν υπάρχει ο απαραίτητος όγκος. Αυτό λοιπόν είναι μία ένδειξη αποτυχίας της αγοράς. Αυτό βλέπουμε ως ένδειξη. Από την άλλη βεβαίως ε, Σωστό είναι να ξαναεξετάζουμε κανονισμούς που είχαν τεθεί ενισχύ πριν από αρκετό καιρό και προψηφιοποίησης ακόμα. και να δούμε αν ταιριάζουν στην εποχή μας. Πρέπει λοιπόν, η σύστασή μας είναι να δούμε ποιες είναι οι αποτυχίες της αγοράς που η παρέμβαση αυτή θα διορθώσει. Όσον αφορά τις κοινωνικές ε, συνθήκες, βεβαίω είναι μια ανησυχία αυτό, έχει τεθεί σε διάφορες πλατφόρμες ε, πριν από λίγες εβδομάδες τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω αν το προσώξατε, υπήρχαν κάποιες ανισχύσεις και απεργίες στη Φιλανδία παραδείγματος χάρη είχαμε απεργία των ταχυδρομείων που οδήγησε σε ε, αλλαγές στο Υπουργείο. Είναι λοιπόν κάτι το πολύ σημαντικό. Και η πρόκληση αυτή υπάρχει. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι η ανταγωνισμού. καθώς η μια πηγή εδώ πέρα είναι, ε, του προβλήματος είναι ότι οι διαφορετικές εταιρείε ε, ε, ακολουθούσαν διαφορετικούς κανόνες. Και βέβαια αυτό στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνήσουμε. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ε, αδειοδότησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες ε, προδιαγραφές. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε 20 λεπτά ε, και θα κάνουμε ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών. Ραντεβού ξανά στις 10. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς με την Κροατική Προεδρία. Ραντεβού στι 10 λοιπόν. So, ladies and gentlemen, please take your seats. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω το δεύτερο μέρος της ε, πρωινής μας ε, συνεδρίασης. Ε, καλωσορίζω την Κορατική Προεδρία που εκπροσωπείται σήμερα από τον κύριο Ιωσίπ Μπίλαβερ, Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και τον κύριο Φράνο Μάτουσιτς ε, από το Υπουργείο Τουρισμού. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Όπως ξέρετε η Επιτροπή μας ε, παρουσίασε τις προτεραιότητες της στην Ολομέλεια και θα τα συζητήσουμε σήμερα με περισσότερες λεπτομέρειες στο μης αρμοδιότητός μας, δηλαδή μεταφορές ε, και τουρισμό. Χαίρομαι για το ότι θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη της ε, ενιαίας ε, ευρωπαϊκής ζώνης μεταφορών των βιώσιμων δραστηριοτήτων και Χαίρομαι ιδιαίτερος για το, οποίο, για το ότι αποδίδεται μεγάλη σημασία στον ε, τουρισμό, κατά το οποίο απασχολεί και την Επιτροπή μας και θα ήθελα ακριβώς ε, να το δούμε πιο συστηματικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνω τώρα να δώσουμε τον λόγο στους δύο υφυπουργούς ε, που θα μιλήσουν 10 λεπτά ο καθένας. Μετά θα ακούσουμε τους συντονιστές, ε, μετά απαντήσεις από τους δύο εκπροσώπους ε, και μετά δίνω τον λόγο στους άλλους ε, βουλευτές. Να δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Μπιλαβέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, Κυρίε και κύριοι βουλευτές, είναι τιμή μου που σας παρουσιάζω σήμερα το πρόγραμμα της Προεδρίας μας στον τομέα των μεταφορών. Γιώση Μπιλάβερ λέγομαι, υφυπουργός ε, θάλασσα μεταφορών και υποδομών. Έχω προετοιμάσει μια παρουσίαση των προτεραιοτήτων μας στην ε, κροατική γλώσσα, οπότε θα ήθελα να μιλήσω τώρα Σας ευχαριστώ. Η Κροατία αναλαμβάνει την ε, Προεδρία σε μια στιγμή μεγάλων προκλήσεων. Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες. Μια Ευρώπη η οποία αναπτύσσεται, ε, η οποία συνδέεται, η οποία προστατεύει και έχει επιρροή. Στην Ευρώπη, η οποία συνδέει, η Προεδρία μας θα δώσει έμφαση στο να ενθαρρύνει πολιτικές ε, οι οποίες θα ενισχύσουν τις διασυνδέσεις εντός της Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα η βελτίωση και η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και δεύτερον ένας ανταγωνιστικός τομέας ε, της ναυτιλίας. Η πρώτη μας ε, προτεραιότητα στις διατροπικές μεταφορές ε, είναι το έξυπνο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών για να απλοποιήσουμε δράσεις που αφορούν την υλοποίηση των δικτύων αυτών. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική προσέγγιση της ε, πρότασης αυτής ε, τον Δεκέμβριο του 2019, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με το Κοινοβουλίο των στομότερο δυνατόν. Και συζητάμε ακόμα τις σχετικές ε, ημερομηνίες. Σκοπεύουμε να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας. Το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη είναι το επόμενο θέμα το οποίο απασχολεί την Προεδρία μας γιατί σχετίζεται με το ΠΔΠ. Βεβαίω ε, αυτό συζητιέται ήδη στην Επιτροπή Ήτρε, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε καθώς έχει μεγάλη σημασία για τις μελλοντικέ επενδύσεις στην προγραμματική περίοδο 2021 2027. Η σημασία δεν αφορά μόνο τις ε, μεταφορές, αλλά και τον τομέα της ενέργειας και τον ψηφιακό τομέα. και αφορά ακριβώς την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε επιτύχει μια συμφωνία κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας ε, το 2019 και όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο να κλείσει τον φάκελο αυτόν. Όσον αφορά την οδηγία για τις συνδυασμένες μεταφορές, η Προεδρία μας ήταν διατεθειμένη να συνεχίσει να εργάζεται επί του θέματος, αλλά υπό το φως των τελευταίων γεγονότων αντιληφθήκαμε πως η Κομισιόν θα αποσύρει το θέμα αυτό και θα το συζητήσουμε αργότερα. Το θέμα για τα δικαιώματα επιβατών σιδηροδρόμων είναι μια βασική προτεραιότητα. Γιατί θα θέλαμε να αυξηθεί η ικανοποίηση των ε, τελικών χρηστών και να προωθηθεί αυτός ο τρόπος μεταφορών που είναι καλός για το περιβάλλον. Το Συμβούλιο έχει φέρει την γενική αυτή προσέγγιση τον Δεκέμβριο του 2019 και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και έχουμε ορίσει τον ε, τριμερή διάλογο για τις 28 Ιανουαρίου. και Βεβαίω στις 11 Δεκεμβρίου η Κορεπέρ επιβεβαίωσε την προσωρινή συμφωνία και αναμένουμε το ίδιο να κάνει και η Επιτροπή σας. Η Κροατική Προεδρία αναμένει την ολοκλήρωση και έγκριση των τριών αυτών θεμάτων την Άνοιξη. Το Συμβούλιο δεν κατάφερε να επιτύχει κάποια συμφωνία για το θέμα της ε, Ευρωβινιέτας και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα οχήματα, δεν ενέκρινε κάποια γενική προσέγγιση το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη που ήθελαν να να δουν τα αποτελέσματα της ε, σχετικής πρότασης για την πρόσβαση στην ε, βιομηχανία και στην αγορά που έδειχναν ε, μια αύξηση των ετοιμάτων για πληροφορίες που ανεβαίνουν στα εθνικά αρχεία. Συνεχίστηκαν και τον Ιανουάριο στο Συμβούλιο οι συζητήσεις όσον αφορά τις αερομεταφορές. Ε, ο φάκελος για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών έχει μπλοκαριστεί εδώ και χρόνια. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Φιλανδίας έγιναν νέα βήματα για να επιταχυνθεί η διαδικασία στα κράτη-μέλη και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και επί Κροατικής Προεδρίας και θα λάβουμε υπόψη την μελέτη για το καθεστώς των ε, δικαιωμάτων αεροπορικών επιφατών. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε κάποια γενική προσέγγιση μέχρι το τέλος της ε, Προεδρίας μας. Όσον αφορά λοιπόν την διαδικασία για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό Σύνδιο, η πρόταση χρονολογείται από το 2013. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει σε αερομεταφορές. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν βεβαίω. Ε, και τα αποτελέσματα στην οικονομία. Εν τω μεταξύ έχει εγκριθεί και ο κανονισμός της ΕΑΖΑ. Το Συμβούλιο Υπουργών ζήτησε από την Κομισιόν το 2018 να εξετάσει το ποιο θα είναι το εύρος των αλλαγών. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς θα αποφύγουμε την συμφόρηση στις μεταφορές και θα μειώσουμε τις ε, εκπομπές. Έχουμε πολλά θέματα, αλλά θα καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για αυτό το ζήτημα. Ε, για να επιτευχθεί κάποια πρόοδος ε, επί της Προεδρίας μας. Η ομάδα εργασίας αερομεταφορών θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά αλλά δεν έχουμε ακόμα κάποιο χρονοδιάγραμμα γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πριν λάβουμε τη νέα πρόταση. Επίσης, προγραμματίζουμε συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής Αερομεταφορών ε, τον Μάρτιο στον Ντουμπρόβνικ. Επιπλέον η Κροατική Προεδρία θα πράξει τα δέοντα για να συνάψει συμφωνίες αερομεταφορών με τρίτες χώρες και ειδικά αυτές οι οποίες έχουν ε, κολλήσει και αφορούν την προετοιμασία του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ. Τώρα, η ναυτιλία. Και η προετοιμασία για την υπουργική δήλωση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ε, των ναυτικών ε, και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ναυτιλίας. Θεωρούμε ότι η δήλωση αυτή είναι μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους ε, για το μέλλον του κλάδου, λαμβάνοντας κατά νου το Green Deal και το ξεκίνημα του νέου νομοθετικού κύκλου. Θα έχουμε κάποιες ε, συναντήσεις 10 και 11 Μαρτίου, ένα άτυπο συμβούλιο στην Απάτια και θα συζητήσουμε με τους ενδιαφερόμενους για τα θέματα αυτά. Θα έχουμε την Υπουργική Διάσκεψη και ελπίζουμε η δήλωση αυτή να μετατραπεί σε συμπεράσματα Συμβουλίου που θα εγκριθούν τον Ιούνιο. Επίσης έχουμε στόχο να μειώσουμε τις εκπομπές ε, αερίου του θερμοκηπίου κατά 50% μέχρι το 2050. Όσον αφορά τις ε, εκδηλώσεις της ε, Προεδρίας μας, θα έχουμε τις ημέρες ε, διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στο ΣΥΒΕΝΙΚ σε συνεργασία με την Κομισιόν και αναμένουμε πάνω από 2.000 συμμετέχοντες. Η ανταγωνιστική και βιώσιμη ναυτιλία λοιπόν είναι μια προτεραιότητά μας και θα έχουμε άτυπο συμβούλιο Υπουργών Ναυτιλίας στην Απατία στις 11 Μαρτίου και την προηγούμενη μέρα θα συναντήσουμε τους ενδιαφερόμενους. Θέλουμε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ναυτική, η ψηφιοποίηση, η ανταγωνιστικότητα και τέλος, στις 29 και 30 Μαρτίου. Θα έχουμε την ε, Σύνοδο Κορυφής Αερομεταφορών στο Ντουμπρόβνικ. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τις δυνατότητες αυτές ε, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και μετά από την παρουσίαση αυτή θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Αναμένουμε λοιπόν διάφορες δυσκολίες, προκλήσεις, πάντα σε πνεύμα διαλόγου. Και ελπίζω να δούμε καλές και συμβαστικές λύσεις. Αυτό και ελπίζω ότι θα έχουμε μια επιτυχή Προεδρία. Πρόεδρο, εμεί ευχαριστούμε κύριε Μπιλαβέρ, ελπίζουμε όλο αυτό το πρόγραμμα που μα παρουσιάσατε θα είναι αντικείμενο προσπαθειών για συμβασμό και τώρα να δώσουμε τη σκητάλη στον κύριο Μάντοσιτ να μα μιλήσει για τον τουρισμό. Ευχαριστώ πρόεδρε, ε, μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, συνάδελφοι, φίλοι. Σήμερα με μεγάλη μου χαρά δράτωμα αυτή τη ευκαιρία να τα συζητήσουμε όσον αφορά τι προτεραιότητε μας για τον ε, τουρισμό κατά την ε, Προεδρία που ασκούμε στο Συμβούλιο. Έχουμε ε, ετοιμάσει ένα ενδελεχές πρόγραμμα, όπω τα είπε ο κύριο Μπιλαβέρ, η Ευρώπη που προστατεύει, που συνδέει, η Ευρώπη που επηρεάζει και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για οριζόντιο τομέα. Γι' αυτό και προτεραιότητες για τον τουρισμό ε, αφορά όλους τους πυλώνες, γιατί ο τουρισμός φέρνει πιο ισορροπή οικονομική ανάπτυξη, συνδέει, συμβάλλει ε, στο να αναβαθμιστεί η φήμη μιας χώρας και βοηθάει στα θέματα ασφαλείας. Ε. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος προορισμός στον κόσμο και είναι σημαντικός παράγων του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 10% από τον τουρισμό, 9% του συνόλου της απασχόλησης στην Ένωση. Και ο διεθνής τουρισμός είναι 6% των εξαγωγών μας και 22% των εξαγωγών υπηρεσιών. Είμαστε τέταρτοι ε, ε, στον τουρισμό μετά από ε, χημικά προϊόντα, αυτοκή και αυτοκίνητα. Και επίσης βοηθά στην προστασία της ε, πολιτικής κληρονομιάς, ε, βοηθά και την αγορά εργασίας αλλά και τις υποδομές αυτά. Αφορούν όλα τα κρατη οπότε θα πρέπει όλα αυτά συστηματικά να τα διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Προεδρία μας θα προωθήσει κάποιες πολιτικές για υπεύθυνο, βιώσιμο τουρισμό αναπτυξιακό και με διαφορετικές ποικίλε ε, πολύμορφες λύσεις σε πολλές ε, περιοχές και θα εστιαστούμε στην συνέργεια με τις ε, τοπικές κοινότητες ανάλογα με την ζήτηση. Θα ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση τεχνολογιών, πληροφοριών, ψηφιακής τεχνολογίας και μια που ο τουρισμός έχει σφαιρικό χαρακτήρα θα πρέπει να αναγνωριστεί περισσότερο μέσα από τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων και πολιτικών. Οπότε θέλουμε να προωθήσουμε τον ε, τουρισμό, ιδίω εκεί που έχουμε υπανάπτυκτες περιοχές, να βοηθήσουμε τη μικροεπιχειρηματικότητα της ΜΜΕ, γιατί έτσι θα έχουμε περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη. Κάποιες ε, δράσεις να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά του τουρισμού και να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε τους προορισμούς. Είναι ο κλάδος ε, ανθεκτικός, βιώσιμος, μακρόπνοα και ωφελεί τις τοπικές ε, κοινότητες. Φέρνει οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική ανάπτυξη στους προορισμούς. Θα προτείνουμε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σήμα, brand, ε, και να προωθήσουμε τον τουρισμό μας σε τρίτες χώρες. Έτσι, με αυτό το μπραντ θα τονίσουμε την υψηλή ποιότητα των προορισμών μας, θα προβάλλεται περισσότερο η Ευρώπη και αυτοί οι προορισμοί. Να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι, να καλύπτουμε την ζήτηση, να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος από την αλλαγή του κλίματος και τις θεομηνίες να προβληθεί περισσότερο η Ευρώπη, πιο αναγνωρίσιμη, παγκόσμια, σταθερός, ασφαλής προορισμός. Αυτά είναι προκλήσεις σημαντικές. Επίσης, ο τουρισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τους θεσμούς για να είναι πιο υπεύθυνος και βιώσιμος. Τέτοια ανάπτυξη να έχει στην Ευρώπη να έχει χαρακτήρα συνεκτικό. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, για να ολοκληρώσω, όσο είχα να σας πω για την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι κάτι που έχει σημασία η οικονομική ανάπτυξη, να είναι υπεύθυνο και βιώσιμος. Να γίνει μια αλλαγή για να κάνουμε την μετάβαση προς μια κοινωνία ουδέτερη περιβαλλοντικά. Επίση, πρέπει να σα πω ότι επανέρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη μου χαρά γιατί είχα διατελέσει παρατηρητή αρχά του 12 μέχρι το 13 πριν δηλαδή γίνουμε πλήρε μέλο γιατί ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσει, τις προενταξιακές τέλο του 11 και γίναμε πλήρε μέρο 4 Ιουλίου του 13 οπότε με χαρά μου επανέρχομαι εδώ και εννοείται ότι σε αυτή τη διαδρομή έχω παρακολουθήσει τις εργασίες της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάτουσιτς για τη συνεισφορά του. Με μεγάλη χαρά σας έχουμε φιλοξενούμενο και εσάς και τον ομόλογό σας. Θα ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις των συντονιστών και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας, για τις μεταφορές. Έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Καλή τύχη για να υλοποιήσετε όλους αυτούς τους στόχους. Δράσεις, πώς να τις πω, που συμπεριλάβατε στο πρόγραμμά σας. Δεν είναι καθόλου εύκολη φάκελη αυτή. Για τα έξυπνα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, έχουμε εισηγηθεί στο ΕΛΚΑ και υποστηρίζουμε πολύ το φάκελο αυτό. Θέλουμε να φτάσουμε σε καλό αποτέλεσμα, αλλά όχι με βάση τη θέση του Συμβουλίου. Έχουν απαλληφθεί πολλά πράγματα από το φάκελο αυτό. Προσπαθήστε να κάνετε ό,τι μπορείτε προς όφελος της ολοκλήρωσης των διαδρόμων αυτών. Ε, γιατί το επιθυμούμε αυτό, την ολοκλήρωσή τους. Για το ΣΕΦ. Ίσως καλό θα ήταν να κάνουμε μια συνεδρίαση. Είμαι εισηγητής για το θέμα του ΣΕΦ για να λύσουμε τα δύο από τα τρία ακόμα εκρεμή θέματα. Για την ε, κατανομή των χρημάτων. Από την, ε, δηλαδή για την πολιτική συνοχής και το θέμα των τρίτων χωρών και να αφήσουμε μόνο ανοιχτό το θέμα του προϋπολογισμού. Αν ψηφίσουμε σήμερα, ο φάκελος θα ξανάρθει στο Κοινοβούλιο ε, και θα είναι ανοιχτός για τροπολογίες. Νομίζω ότι θα χρειαστούν να κάνουμε και άλλα πράγματα στο Κοινοβούλιο, να, κάνουμε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα. Για τα δικαιώματα των επιβατών έχετε ασχοληθεί ήδη με αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως να ανοίξετε τώρα τη συζήτηση η οποία έχει μπλοκάρει το και μεγάλο χρονικό διάστημα για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, χωρίς κανέναν λόγο. Είναι δύσκολο ο φάκελο, αλήθεια είναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Ίσως θα μπορούσατε να κοιτάξετε λιγάκι και τα σλότ, τις χρονικές θηρίδες. Δεν είναι στο πρόγραμμά σας, αλλά ο κλάδος περιμένει αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό. Μα είπε θα κάνετε πολλές προσπάθειες. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε όμως ε, λίγο περισσότερα για διάφορους φακέλους που τους αναφέρατε πολύ χοντρικά. Λοιπόν, για τον τουρισμό. Ακόμα ασχολούμαστε με το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Ίσως πείσετε τελικά τα κράτη-μέλη να βάλουν χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για τον τουρισμό. Το Κοινοβούλιο θα σε υποστηρίξει. Ο κύριο Μαρινέσκου. Και τώρα... Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινέσκου και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Ντάνιελσον από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ και του δύο υπουργού που ήρθαν εδώ και που μα παρουσίασαν τι προτεραιότητε για του επόμενου 6 μήνε. Είμαι ιδιαίτερο ε, ικανοποιημένο με τι φιλοδοξίε σα για τον τομέα των μεταφορών. Ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να τα καταφέρετε να υλοποιήσετε του περισσότερου στόχου. Φυσικά το Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το δίκτυο των διευρωπαϊκών δικτύων, το TEN-T, δίκτυα μεταφορών. Είναι σημαντικό για τις α, επενδύσεις των μεταφορ, ε, στις υποδομές αυτές. Ε, και είναι πολύ σημαντικός ο, στόχος αυτός για να υλοποιήσουμε τις α, κλιματικές υποχρεώσεις μας. Για το, τις πολύτροπες μεταφορές. Εμείς ως σοσιαλιστές πιστεύουμε ότι είναι λάθος της Κομισιόν να αποσύρει την πρόταση από τις ε, συνδυασμένες μεταφορές. Εμείς θέλουμε να πάμε σε τριμερή διάλογο ε, μαζί σας. Αν μπορούμε να πείσουμε την Κομισιόν να το ξανασκεφτεί το θέμα και να μην το αποσύρει, εμείς θα ήμασταν ικανοποιημένοι να διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο ως Κοινοβούλιο και να κλείσουμε το θέμα αυτό πριν το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε άλλα δύο χρόνια, ούτως ώστε να έχουμε πιο φιλόδοξη πρόταση. Νομίζω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις τους μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή τη φιλοδοξία ε, και να τα καταφέρουμε πριν το καλοκαίρι. Κατάλαβα ότι δίνεται προτεραιότητα στις τελικές διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, σαφείς ε, ευρωπαϊκοί κανόνες και εγγύησεις για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων, ε, ειδικά όταν, ε, αν θέλουμε να πείσουμε τους επιβάτες να αφήσουν άλλες, άλλα είδη μεταφορών και να πάνε στο σιδηρόδρομο. Επίσης, το θέμα της αεροπορίας. Είχα καταλάβει ότι είναι προτεραιότητά σας ε, το να ξεμπλοκάρετε κάποιοι, κάποιους φακέλους που ήταν μπλοκαρισμένοι εδώ και χρόνια. Θα το ήθελε πάρα πολύ αυτό το κοινοβούλιο και κυρίως οι σοσιαλιστές. Γιατί οι αερομεταφορές ε, είναι ένα τομέα όπου σε ό,τι αφορά την νομοθεσία που τον διέπει, καθυστερούμε. Ίσως κάτι ξέχασα, έχασα από αυτά που είπατε. Θα μπορούσατε να μα εξηγήσετε πιο συγκεκριμένα πώς θα προσπαθήσετε να ξανανοίξετε τι διαπραγματεύσεις για αυτό το φάκελο και να ξεμπλοκάρετε το θέμα αυτό και ποιο είναι ο χρονικός ορίζοντας ε, θεωρείτε για να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα στα θέματα της αεροπορίας. Προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία μαζί σας τους επόμενους μήνες. Συμφωνώ και με τον Μαρινέσκου για το θέμα του τουρισμού. Αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια γραμμή προϋπολογισμού για τον τουρισμό θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Αυτό το βλέπουμε πολύ καλό μάτι αυτή η Επιτροπή και όλο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Ναχταρά από το Ρινιού. Καλωσορίζω τους Υπουργούς. Καλή αρχή κάνει η Προεδρία το 2020 και εστιάζει σε πολλά και διάφορα θέματα. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ας πούμε, τα δικαιώματα των επιβατών αερομεταφορών, αλλά ακόμα έχουμε ακόμα μια νέα χρονιά και δεν έχουμε ακόμα τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Το ανέφεραν και άλλοι συναδελφοί. Το θέμα της αεροπορίας, πολύ σημαντικό. Αλλά ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι τόσο σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερες καθυστερήσεις, ε, σε λιγότερες αλλαγές της διαδρομής των αεροπλάνων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 10% μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, το πιο σημαντικό από όλα. Το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο ε, λήφθησαν ε, αποφάσεις για κανονιστικά θέματα. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το πώς εσείς θα προχωρήσετε για να τελεσφορήσει αυτός ο φάκελος ε, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλο χρόνο εξάλλου μπροστά μας. Από τους πράσινους, ο κύριος Κάφ. Να συνεχίσω. Στο θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Θέλουμε εναέριες οδούς που να είναι πιο άμεσες. Θέλουμε εξοικονομήσεις που θα προκύψουν ακριβώς από αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν ε, διευκολύνουμε τις αερομεταφορές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πετάνε. Και σε ένα κόσμο που έχουμε θέμα ε, με, τις, με τους στόχους μας για το διοξίδιο του άνθρακα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τι προσπάθειες μπορούμε να κάνουμε ή θέλετε να κάνετε, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε δεν υπάρχει αύξηση στις εκπομπές από την αεροπορία, εάν ε, υλοποιήσουμε το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμπομινώση από το ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Υπουργοί, από, τους, από την Κροατία. Σας καλωσορίζω. Συχνά σε αυτήν την Επιτροπή, όπως ξέρετε, οι αντιθέσεις δεν είναι μεταξύ αριστεράς ε, και δεξιάς, αλλά ανάμεσα συμφέροντα των χωρών της ε, Δύσης και της Ανατολής. Παραδείγματο χάρη, είχαμε μια σκληρή διαπραγμάτευση στο θέμα της κινητικότητας, όταν το διπραγματευτήκαμε αυτό το πακέτο, και η Κροατία θα μπορούσε να βοηθήσει για να ξεπεράσουμε αυτή, αυτό το ρήγμα, λόγω της θέσης της, της ιστορίας της κτλ. Αυτή την ε, αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης. Πολύ σύντομη παρέμβαση. Για τον Μπρένερο έχουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε τα συμφέροντα θεμητά της Αυστρίας. Αλλά όσο δεν θα έχουμε το σιδηροδρομικό αυτό τούνελ για να μειωθεί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αυστρίας, οι περιορισμοί που υπήρχαν ήδη και που αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο και που ε, ανησυχούν και τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, έχουμε διάλογο δηλαδή με τις εμπλεκόμενες περιφέρειες Νομίζω ότι όσο δεν λυθεί αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να ε, εξεταστεί πάρα αυτά. Έχω γράψει μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του Μπρένερο, για να βρεθεί μια λύση. Για να εγγυηθεί τα συμφέροντα όλων. Γιατί δεν θέλω εδώ πέρα να σας αναφέρω το, την ελεύθερη κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα εμείς, αλλά καταλαβαίνω και το πρόβλημα της Αυστρίας. Θέλουμε απλώς να, να κυκλοφορούν όσοι πρέπει να κυκλοφορούν, εύκολα. Κάτι άλλο, πολύ γρήγορα. Μερικές φορές υπάρχει ε, ολιγοπόλιο στις ναυτιλιακές εταιρείε. Έχουμε κάποιες ναυτιλιακές που γίνονται και τερματικοί σταθμοί, που κρατούν, έχουν στα χέρια τους όλες τις θέσεις του κλάδου. Θέλω να βάλετε Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέους κανόνες για να εξασφαλίσετε την, τον ανταγωνισμό και την δυνατότητα να μπαίνουν πολλές εταιρείε ε, και να παρέχουν υπηρεσίες. Δεν θέλουμε ολιγοπόλια γιατί αλλιώς θα έχουμε στρεβλώσεις ε, του ανταγωνισμού στα λιμάνια μας. Από το ECR θα πάρει κάποιος το λόγο. Κύριος Βός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο πράγματα να πω. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις σύντομες πτήσεις εντός της ε, Ευρώπης, τότε θα πρέπει ο χρόνος ε, ταξιδιού και το κόστος ε, των διεθνών τρένων να μειωθεί. Αυτό βεβαίως απαιτεί συνδέσεις στο σύστημα και μεταξύ κρατών μελών. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αρκετά και είναι μια στενοπός που πρέπει να ξεπεραστεί. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η εσωτερική ναυτιλία και η ακτοπλοεία σε σχέση με το Green Deal. Μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις που κάνουν τεράστιες ε, επενδύσεις, πολύ μακροχρόνιες και πρέπει να μπορούν να τις αποσβέσουν. Όσο πιο καθαρές ε, τόσο το καλύτερο, αλλά πρέπει να έχουν και χρόνο ε, Οπότε θα πρέπει το Green Deal να μην τους ε, κόψει τα πόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα για την ΚΟΕ η κυρία Κουντουρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίλαβερ και τον κύριο Μάτουσιτς για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της κρατικής προεδρίας Σχετικά με την πολιτική μεταφορών, το πρόγραμμα της Προεδρίας φαίνεται να μας ικανοποιεί, καθώς και μετά την υιοθέτηση από την Επιτροπή του Green Deal, θα ξεκινήσει πολύ σημαντική συζήτηση για τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας και της αεροπορίας και θα πρέπει βέβαια στόχος των συζητήσεων αυτών να είναι οι δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο θέμα της νησιωτικότητας. Ε, κύριε Μπίλαβερ, ε, η Κροατία όπως και η Ελλάδα Έχουμε πάρα πολλά νησιά. Είναι σημαντικό λοιπόν τα νησιωτικά κράτη να προβάλλουν τις ανάγκες της νησιωτικότητας γιατί δεν είναι για όλους αυτονόητα. Ειδικά το ζήτημα των μεταφορών είναι ζωτική σημασία για την νησιωτικότητα και οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ δύσκολες λόγω του αυξημένου κόστους μεταφορών, μεταφορικών σε ενέργεια, τρόφιμα, ακόμα και νερό αλλά και τα απορρίμματα. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει αυτή την κατάσταση και πρέπει να λάβουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό ζήτημα που είναι ήδη οξύ και έχει και γεωστρατηγική σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να αναδείξετε αυτές τις ειδικέ ανάγκες της νησιωτικότητας και πώς θα τις εντάξετε στις διεργασίες της Προεδρίας σας τους επόμενους έξι μήνες. Ε, στο φίλο μου τον Φράνο Μάτουσιτς ε, θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήμουν βέβαιη ότι στο πρόγραμμα θα υπάρχει ο τουρισμός. Είναι γνωστό ότι είναι τομέας καταλήτης για την ανάπτυξη της οικονομίας και συνολικά ε, προσφέρει διέξοδο σε περιοχές και με μειωμένες κατά τα άλλα οικονομικές δυνατότητες, αλλά ε, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ε, πραγματικά έχει τη δυνατότητα να δώσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην οικονομία του κάθε κράτους και φυσικά της Ευρώπης που όπως πολύ σωστά είπατε είναι το 10% του ΑΕΠ και η Ευρώπη είναι ο πρώτος μεγάλος προορισμός. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξετε αυτό που ανέφεραν και οι συνάδελφοι ε, το κομμάτι που αφορά τον προϋπολογισμό. Ε, έχουμε κάνει ένα αίτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για ένα συμβολικό ποσό των 300 εκατομμυρίων για την περίοδο 2021-2027 και πρέπει να πιστούν όλοι και οι συναδελφοί σας και το Συμβούλιο για το δίκαιο αυτό αίτημα. Τέλος, θα ήθελα να μελετήσετε και το ψήφισμα για την Thomas Cook, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό ψήφισμα που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί για μα είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να δημιουργηθεί αυτό ο ευρωπαϊκό μηχανισμό για τη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό, πράγμα το οποίο δεν αντιλαμβάνονται όλοι. Ε, και τι εννοούμε. Ένα μηχανισμό ο οποίο θα παρέχει υποστήριξη στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν κοινέ προκλήσει, όπω είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω τη κλιματική αλλαγή, θέματα ασφάλειας, ζητήματα ασφάλειας, το προσφυγικό, ο υπερτουρισμός, η υπεύθυνη ε, βιωσιμότητα και όλες αυτές οι, οι προκλήσεις βρίσκονται και στο πρόγραμμα της δικής σας Προεδρίας. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να το μελετήσουμε και να αναδειχθεί ε, το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. And ε, τώρα, λέει ο Πρόεδρος, Πάμε στις ε, απαντήσεις. Ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος? Ο κύριος Μπιλαβέρ. Στα κροατικά. Ναι, να σας απαντήσω εγώ πρώτος και σας ευχαριστούμε για αυτές τις επικοδομητικές, τις εύστοκες ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθήσατε αυτά που σας παρουσιάσαμε. Έχουμε ένα σωρό ερωτήσεις, τις πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα-πρώτα ε, για τον κύριο Μαρινέσκου. Ναι, λαμβάνω υπόψη αυτό το οποίο είπατε ήδη, τα έχουμε πει επανειλημμένα. Και αναφερθήκατε στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Είπαμε στην εισήγησή μας ότι για μας ε, είναι μια προτεραιότητα στην ομάδα για τις ε, ε, συνδυασμένες μεταφορές. Και ο, ήδη από νωρίς ξεκινήσαμε την ανάπτυξη υποδομών στους βασικούς ε, διαδρόμους και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία το 2030. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να κάνουν ό,τι μπορούν για τον σχετικό κανονισμό. Αυτόν που θα διέπει ε, τις ευφύ συνδυασμένες μεταφορές. Γίνονται συζητήσει για το πότε θα αρχίσουν οι πράγματα στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε αυτό να γίνει όσο γίνεται συντομότερα για να ξεκινήσουν τριμερεί διάλογοι. Τώρα, όσον αφορά τι συγκοινωνίε. Μια σειρά βουλευτών αναφερθήκαν σε αυτό στο θέμα των μεταφορών. Έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Ουρανό και έχουμε επίση και τα δικαιώματα των ε, επιβατών όσον αφορά τις αερομεταφορές. Δεν θέλω τώρα να κάνω κάποιες κούφιες υποσχέσεις, ούτε μπορώ να πω ε, έτσι κάποιες ημερομηνίε που ενδεχομένω δεν ισχύουν, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Αλλά αυτό το πρόβλημα εκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια και θέλουμε κάτι να κάνουμε. Αν λύσουμε αυτά τα ζητήματα, τότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας βοηθήσετε κι εσείς. Αλλά βέβαια το πρώτο βήμα πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ε, Δεκέμβριο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, ποικίλες απόψεις στο Συμβούλιο και διαφορετικές. Γι' αυτό και εμείς παρουσιάσαμε στην Επιτροπή τις προτεραιότητές μας και ζητήσαμε να γίνει μια επαναξιολόγηση. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν ανάγεται στο 2013. Επίσης θα γνωρίζετε ότι έχει αυξηθεί ε, ο όγκος των αερομεταφορών, ότι έχει εξελιχθεί επίσης και η τεχνολογία και συνεχίζει και εξελίσσεται με ταχύτητα ρυθμούς και έχουμε πάρα πολλές εκπομπές. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Πάντως, μας ικανοποιεί πάρα πολύ η πρόταση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία. Πρόκειται για μια συμφωνία που θα έχει επιπτώσεις στις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και τις σιδηροδρομικές διότι θέλουμε να υπάρξει μετακίνηση των μεταφορών προς σιδηρόδρομο και εσωτερικές πλωτές οδούς. πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες προτάσεις, να αρχίσουμε τις επαφές εμείς με τα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι θα σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος που χρειάζεται να γίνει. Σε σχέση με τα υπόλοιπα που ρωτήσατε, ο κ. Καμπομπανέζε μας είπε για το Μπρένερ και την ορεινή διάβασή του. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Θα πρέπει εκεί να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος. Όμως υπάρχουν εμπορικές ανάγκες και διάφορα ζητήματα με τις τοπικές κοινότητες. Αυτά δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Μπορώ να σας πω ότι στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας είμαστε κράτος μέλος και αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με τις ε, γειτονικές μας χώρες. Πάντα αναζητούμε λύσεις συμβαστικές. Πάντως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι σαφές ότι αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται όσο γίνεται καλύτερα. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα πνεύμα καλής γειτονίας και έτσι να γίνεται προσπάθεια αναζήτησης λύσεων. Ε, βέβαια και εμείς είμαστε πρόθυμοι προς τούτο και θεωρούμε ότι όλα αυτά βοηθάνε, σας το λέω από την εμπειρία μου. Ο κύριος επίσης ανέφερε και εκείνος για την Πράσινη Συμφωνία Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα προβλήματα. Παγκοσμίω διαπιστώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η Ευρώπη επίσης έχει πληγεί από τέτοια φαινόμενα. Εμείς έχουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη χώρα μας, ε, επίσης ε, ξηρασία το καλοκαίρι, τα έχετε διαπιστώσει και γνωρίζεται και για τις πυρκαγιές στην Αυστραλία αλλά και τις πλημμύρες στον Καναδά. Είναι κοινό συμφέρον μας να βρεθούν κάποιες λύσεις. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωτοπόρα και να λάβει την πρωτοβουλία για κάποιες ε, αλλαγές που θα γίνουν όχι μόνο εδώ αλλά σε όλο τον κόσμο και εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Εμεί να ξεκινήσουμε τι αλλαγέ που χρειάζονται και αυτό να γίνει το του δυνατόν. Γιατί ο χρόνο πιέζει. Πάρα πολύ θετική η πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία. Ήδη υπάρχουν επιπτώσεις στις μεταφορές γιατί γνωρίζουμε ε, το θέμα των ε, εκπομπών από τις ε, μεταφορές. Όλες τις μεταφορές. Και αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. για όσον αφορά τις εμπορικές μεταφορές, τη μετακίνηση αυτών των μεταφορών από το δρόμο, στο σιδηρόδρομο και στις εσωτερικές πλώτες όδους και θα πρέπει όλα αυτά να τα καλύψουμε με το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και έτσι να δοθεί πρικοδότηση σε αυτές τις ε, μεταφορές που θέλουμε να τονώσουμε. Τώρα, για τα γιοταχή αυτοκίνητα. Θα πρέπει και εδώ να γίνει μια αλλαγή. Αλλαγή στα καύσιμα. Θα πρέπει οι χώρες σας να κάνουν μια τέτοια αλλαγή. Επίσης, στην Οπάτια έχουμε αυτή την διάσκεψη για τις θαλάσσιες μεταφορές. Παρακαλώ τα κράτη-μέλη να προσυπογράψουν το σχετικό έγγραφο. Αυτό το έγγραφο θα ενσωματωθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θέλουμε οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη να ε, προχωρήσουν, να αποκτήσει η Ευρώπη ανταγωνιστικότητα πέραν του θέματος της ε, μείωσης των εκπομπών. Μείωση εκπομπών επομένω θέλουμε, θέλουμε ψηφιακή τεχνολογία, θέλουμε καινοτομία στον κλάδο αυτό και έχουμε υποσχεθεί να δουλέψουμε προς αυτό το μέτωπο και ελπίζουμε ότι η σχετική διακήρυξη, η τελική δήλωση τέλος πάντων στη Σοπάτια να εγκριθεί. Κυρία Κουντουρά, είστε Ελληνίδα και μας αναφέρατε για το πόσο χρειάζεται να υπάρξει επικοινωνία και διασύνδεση των νησιών. Και εμείς στην Κροατία έχουμε πολλά νησιά, έχουμε πάνω από χίλια νησιά και ξέρουμε καλά το πρόβλημα της επικοινωνίας και διασύνδεσης των ε, νησιών και γνωρίζουμε ότι έχετε τη σχετική εμπειρία αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και η Ισπανία. Όλοι θέλουμε να διατηρηθούν ε, οι τοπικές κοινότητες στα νησιά, μην υπάρχει δημογραφική συρρήγνωση θέλουμε, αντίθετα να αναπτυχθούν αυτές οι κοινότητες να μεγαλώσουν και επίση θέλουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές ε, και αυτές οι υποδομές να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να υπάρχουν υψηλά στάνταρ όσον αφορά τις επενδύσεις, να προστατευτεί το περιβάλλον και να υπάρχει βιωσιμότητα. να χρησιμοποιηθεί από τους μεταφορές ε, μια εναλλακτική ενέργεια όπως το υδρογόνο ή ο, ηλεκτρο, ο ηλεκτρισμός. Εμείς έχουμε αναπτύξει στην Κροατία την ιδέα του έξυπνου εφιούς νησιού, Smart Islands, ε, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τα είδη διατροφής και τις βιώσιμες μεταφορές. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε μια ε, υποδειγματική εφαρμογή για να αναπτύξουμε τα νησιά μας, να σταματήσουμε την μετανάστευση από τα νησιά, να κρατήσουμε κυρίως τους νέους στα νησιά. Γιατί ναι, έχουν εκεί οικογένειες, αλλά βέβαια χρειάζεται να τους δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης εκεί. Α, και κάτι άλλο. Όταν μιλούμε για αερομεταφορές και είχαμε πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό, μια σειρά από βουλευτές ασχολήθηκαν με το θέμα, το οποίο είναι βέβαια σημαντικό και μας κάνει να προσπαθήσουμε σε αυτό το μέτωπο στο εξάμεινό μας. Θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι και στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας γίνανε κάποια πράγματα. Εμεί αυτά θα τα κρατήσουμε, θα τα σεβαστούμε και τι θα θέλαμε να κάνουμε. Θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη τη μελέτη της Κομισιόν όσον αφορά ε, τα θέματα των επιβατών των αερομεταφορών. Και με βάση αυτή τη μελέτη κάνουμε επαφές με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές λύσεις, να τις κατεβάσουμε στο Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι τελικά θα σημειωθεί κάποια πρόοδος. Πρόοδος σημαντική και θέλουμε να υπάρχει σφαιρική προσέγγιση. Όσο γίνεται. Ξέρω ότι ο κύριος Μανέσκο προσπαθεί. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ο πρόεδρος. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου, την κυρία Κοντουρά και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις που μου έθεσαν. Υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή, ένα νήμα που μας καθοδηγεί, που είναι το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να δοθούν συγκεκριμένα μέσα, συγκεκριμένοι πόροι στον ε, τουρισμό. Το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε μια τέτοια πρόταση, πρότεινε να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες υποστήριξης των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων στον, τομέα του τουρισμού μέσω των προγραμμάτων της ενιαίας αγοράς. Έτσι έχει η κατάσταση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού για τον τουρισμό. Περιμένουμε στις 27 και 28 Απριλίου στον Ντουμπρόβνικ να γίνει μια συζήτηση στην Σύνοδο Κορυφής που θα διοργανώσουμε και όλοι οι Υπουργοί Τουρισμού θα παραστούν, φαντάζομαι. Και ακριβώς λοιπόν εκεί θα τους υποβάλουμε το ερώτημα πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τον τουρισμό, πώς μπορούμε να το εξασφαλίσουμε μια καλύτερη θέση. Προφανώς. Μαζί με την κυρία Κουντουρά είχα πολλές συζητήσεις σε διάφορες φάσεις, σε διάφορα βήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Κουντουρά για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση για τον τουρισμό, ιδίω τις δυνατότητες που έχουμε να αναπτύξουμε τις ε, περιοχές της Υπέθρου που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά. Ακριβώς γι' αυτό ε, συμμετείχαμε σε πολλές κοινέ πρωτοβουλίες και είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιαστούν στα τέλη Απριλίου πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες και θα συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα που θα υιοθετηθούν τελικά το Μάιο. Συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα γίνει πολύ ενδελεχή συζήτηση για το θέμα του τουρισμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των περιοχών τη Υπέθρου και για την εξασφάλιση ενό συνδέσμου ε, με το γεωργικό κλάδο, την ανάπτυξη της ζήτησης στις περιοχές αυτές και της ε, τουριστικής ζήτησης, όχι μόνο γενικά της ζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός. Είναι μία από τις πιο σημαντικές ε, επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Επίσης, κάτι άλλο που είναι σημαντικό, και εδώ θέλω να μιλήσω λιγάκι για την κροατική περίπτωση ότι ο τουρισμός είναι το 20% του ΑΕΠ μας. Και για όλα τα κράτη-μέλη, ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς τώρα που έχουμε ανάγκη. Το Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία του θέματος. Ας πούμε, πολύ σημαντική είναι η περίπτωση Thomas Cook. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μηχανισμούς οι οποίοι μας επιτρέπουν να αντιδρούμε ε, παρκώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Είτε στον τομέα των μεταφορών, είτε σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, είτε σε περίπτωση που έχουμε μετρολογικές ε, καταστροφές, ας πούμε, που, επιτρέπ, που επηρεάζουν τις ε, μεταφορές και επηρεάζουν τελικά και τον τουρισμό. Είναι σημαντικό να αντιδρούμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ε, παίζονται εδώ πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Στην περίπτωση της Κροατίας, ο τουρισμός ε, αναπτύσσεται κυρίως στα νησιά. Και εκεί βλέπουμε την ανάγκη να συνδέουμε καλύτερα τα νησιά, ούτως ώστε οι επιβάτες να πηγαίνουν το χρονικό δυνατόν στα νησιά, να μην χάνουν χρόνο αλλού, για να γίνουν πραγματικά πιο ελκυστικοί αυτοί οι προορισμοί. και για να εξασφαλίσουμε τη ζήτηση πέρα από την πολύ στενή έντονη τουριστική περίοδο να ζητήσουμε δηλαδή, να εξασφαλίσουμε δηλαδή μια μόνιμη ζήτηση. Για μας είναι πολύ σημαντικό οι τοπικές κοινότητες να ικανοποιούνται από, τα, από τους καρπούς του τουρισμού και να επιτρέπει ο τουρισμός στις ε, κοινότητες αυτές να αναπτυχθούν και να κατανέμουν καλύτερα τους καρπούς του τουρισμού και να μπορέσουν τελικά να παίρνουν κάποιες αποφάσεις πιο αυτόνομα για την ανάπτυξη της προσφοράς ε, μαζί με τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, συχνά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά για να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο σε, στις τοπικές αυτές κοινότητες. Σας ευχαριστώ όλους, αλλά ιδιαίτερα στην κυρία Κουντουρά που είναι φίλη και συνάδελφος εδώ και πολλά χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του τουρισμού. Ευχαριστώ. Πρώτος γύρος. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Για το δεύτερο γύρο θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά σε κάθε έναν από τους ευρωβουλευτές για να κάνει σχόλιο ή ερώτηση. Ο κύριος Ντελή είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ την κρατική Προεδρία που ήρθε εδώ. Η πολιτική διεύρυνση διεύρυνσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Προεδρίας σας. Ε, το Μάιο θα γίνει μια σύνδοση κορυφής που θα είναι ας πούμε η κορονίδα της προσπάθειάς σας. Νομίζω ότι πρέπει να, βάλετε να λάβετε υπόψη τις απόψεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ό,τι αφορά ειδικά τις πολιτικές μεταφορών. Θα χρησιμοποιήσετε την ε, προσφάτως δημιουργηθήσα Επιτροπή Μεταφορών που είναι μια κοινή προσπάθεια της Κομισιόν και των χωρών αυτών, των Δυτικών Βαλκανίων δηλαδή. Ε, επίσης, η διασυνοριακή συμφόρηση. Και δεν μιλάω για τις υποδομές ε, και τη σύνδεση που έχουμε με αυτές τις χώρες, γιατί είσαστε γείτονα ε, με αυτές τις χώρες, με κάποιες από αυτές τις χώρες, όπως και η χώρα μου. Ε, όπως και χώρα μου. Αλλά κοιτά, μιλάω κυρίως για τα τελωνία και τις τελωνιακές ε, διαδικασίες, γιατί συχνά το καλοκαίρι βλέπουμε χιλιόμετρα ουράς φορτηγών στα σύνορα, να συνοθούνται στα σύνορα. Κάτι που δημιουργεί πάρα πολλέ εκπομπές, δημιουργεί καθυστερήσει και φυσικά δεν είναι ανθρώπινε συνθήκες ε, εργασία για τους οδηγούς. Και ούτε βοηθάμε έτσι στην υλοποίηση των στόχων της ε, Πράσινης Συμφωνίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα αυτό των τελωνιακών διαδικασιών στα σύνορα. Ευχαριστώ κύριε Ντελή. Φλέγκορ. Και μετά οι επόμενοι ομιλητές. Εγώ, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω κι εγώ. Και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Κροατική Προεδρία. Μια συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, κύριε και μια ερώτηση. Ακούσαμε πολλά για το συνδέοντας ε, την Ευρώπη αλλά και τις διασυνδέσεις γενικά και είναι θέμα ισότητας. Ε. Η Ανατολική Ευρώπη ιστερεί και αυτό είναι ευδιάκριτο ε, ειδικά η κατάσταση στις μεταφορές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές και πόσο διαφέρει η Ανατολική από τη Δυτική Ευρώπη ας πούμε, το πρώτο νυχτερινό τρένο από την Βιέννα στις Βρυξέλλες, ε, από τη Βιέννη στις Βρυξέλλες ξεκίνησε χθε. Αυτό για μας μοιάζει με διαστημικό ταξίδι. Δηλαδή από την Πούλα στη Βουδαπέστη χρειαζόμαστε 5,5 ώρες. Ε, ε, φαντάζεστε άρα την ταχύτητα για την οποία μιλάμε. Είναι όμως ε, σημαντικό να πούμε ότι για τους λόγους αυτούς οι ταξιδιώτες όταν έχουν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι τελικά θα πάρουν το αυτοκίνητο και βεβαίω ε, αυτά δεν είναι καλά για το περιβάλλον, είναι και πιο ακριβά και ακούσαμε επίσης χτες τα στατιστικά στοιχεία για την εθνισιμότητα στους δρόμους και βεβαίως πρώτη στον κατάλογο είναι η Ανατολική Ευρώπη. Όταν λοιπόν θα αναθεωρήσουμε τους ευρωπαϊκούς ε, διαδρόμους ε, μεταφορών σας παρακαλώ να δράσετε εγκαίρως για να μην χάσουμε χρόνο. Και μια που λέτε ότι αναμένετε το Green Deal. Η Κροατία έχει μόλις 1,3% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι η προτελευταία στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι πώς θα φτάσουμε το 14% το 2030 που είναι ο στόχος. Κύριε Μάτουσιτς, έχω δύο προτάσεις. Πρώτον, η πρώτη σχετίζεται με το ότι είχαμε εδώ πριν από δύο μήνες μια μελέτη για τον υπερτουρισμό. Δεν θα μπω τώρα στο θέμα αυτό, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερες ε, πόλεις στην Κροατία και στην Ευρώπη. Μας ε, μίλησαν και οι συναδελφοί μας από το Λονδίνο, ότι αυτοί που εργάζονται στο Λονδίνο στις ε, δημόσιες ε, υπηρεσίες ε, πληρώνονται ένα επιμίσθιο λόγω του κόστους ζωής στο Λονδίνο. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε το ΠΔΛΤΑΠ να κάνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση και τέλος όσον αφορά τους επισκέπτες μας από μακρινές χώρες πώς θα μπορούσαμε να τους συνδέσουμε καλύτερα με κοινέ διαδρομές στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Μοντέρο Ντεγκιλέρ και μετά στον κύριο Ερτούγ. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τους δύο υπουργούς επίσης να τους ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε που ήρθανε, τους ευχαριστούμε που μας ε, εξήγηλαν το πρόγραμμα εργασίας και θέλω να σας ευχηθώ ολόθερμα καλή επιτυχία. Μας μιλήσατε για τις μεταφορές, μας μιλήσατε για τις ε, υποδομές, ε, για τις θαλάσσιες μεταφορές, για τον τουρισμό. Χρειάζονται πάντως συγκεκριμένες δράσεις. Γι' αυτό και εγώ θέλω να χτυπήσω ένα καμπανάκι όσον αφορά τα νησιά, όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει ένα νομικό θέμα, υπάρχει μία διάταξη για την απότερη περιφέρεια στις ε, συνθήκες και αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Έχουμε τώρα την φιλοδοξία ε, της Πράσινης Συμφωνίας, οπότε θα πρέπει και από τον κλάδο του τουρισμού να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες αυτών των νησιών, αυτών των ε, απότερων, όπως λέμε, περιφερειών που αφορά τρία κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε για το όσο μας εξηγήσατε στην αρχή που μας είπατε ε, πόσο οριζόντιο χαρακτήρα έχει ο τουρισμός, πόσο σημαντικός είναι για κάθε κλάδο της οικονομίας. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία, τα είπαμε αυτά. Κάναμε συζητήσεις, κάναμε ε, ψηφίσματα για διάφορους στόχους, θέλουμε να έχουμε βιώσιμο τουρισμό και για αυτό το λόγο χρειάζονται κονδύλια. Τα είπε αυτά το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα και μιλήσαμε για 300 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπήρξε κάποια απάντηση, κάποια ανταπόκριση. Τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνετε για αυτό το κονδύλιο, τι θα γίνει από το Συμβούλιο στο επόμενο πολιετές χρηματοοικονομικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ε, θα πρέπει να κάνετε μια τέτοια δέσμευση και με τα διαρθρωτικά ταμεία και με τέτοια κονδύλια να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για βιώσιμο τουρισμό, για ασφάλεια, για να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή και τις ΜΜΕ. Ξέρουμε ότι περισσότερες επιχειρήσεις του τουρισμού είναι ΜΜΕ. Μιλήσατε και για τις κρουαζιέρες, για τις θαλάσσιες μεταφορές. Όλα αυτά είπατε συνολικά θα τα διεκπεριώσετε. Επίσης, ε, μια task force θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα αυτό, να γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες. Παρακαλώ, κάντε μια προσπάθεια απευθυνθείτε στην Κομισιόν να κατεβάσει μια νομοθετική πρόταση η Κομισιόν, ούτω ώστε να υπάρξει αυτό το κονδύλιο. Έχουμε κάνει μια τέτοια προσπάθεια εδώ και κάποια χρόνια να αντικατοπτρίζονται οι ανάγκες ε, στις προτεραιότητες και στον προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένως να μπορέσει να βοηθήσει. To Mr. and then to Mr. Newton Ευχαριστούμε. Ο επόμενος, ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σερτούγ. Καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Εύχομαι επιτυχή Προεδρία και μπορείτε να βασιστείτε στην στήριξή μας για τις προοδευτικές πολιτικές σας. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της αεροπορίας γιατί η απάντησή σας ήταν μακροσκελής αλλά δεν περιείχε πολλή ουσία. Θα να γνωρίζω λοιπόν τι μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά τις διαφορετικές ε, συμφωνίες. Θα τις οριστικοποιήσουμε. Έχετε κάποια στρατηγική για το πώς θα πείστε τα κράτη-μέλη που κυρίως επιβραδύνουν την διαδικασία. Αυτό θα μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ερτούγ. Τώρα κύριος Νιούτον Ντάν ε, και κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Προεδρία. Έχω να κάνω μια ερώτηση για την διαδικασία στο Συμβούλιο. Όλοι γνωρίζουμε το ότι το Κοινοβούλιο είναι η εκπρόσωποι του λαού. Συνεδριάζουμε δημοσίω, μπορούν να μας ακούσουν, μπορείτε εσείς να έρθετε να μας ακούσετε. Δημοσιεύουμε τα πάντα, τα πρακτικά, στο site κτλ. Το Συμβούλιο όμως όχι. Είναι μυστικοπαθές. Εάν θέλουμε λοιπόν να μας ακολουθήσουν οι λαοί της Ευρώπης και να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Βρετανός που πληρώνουμε υψηλό τίμημα γιατί δεν έχει συμβεί αυτό στη χώρα μας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημοσίως θα επιτρέψετε στους πάντες να γνωρίζουν το τι συμβαίνει εκεί μέσα γιατί δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση αυτή τη στιγμή θα γνωρίζει το κοινό εάν υπήρξε ε, ψηφοφορία ή έγινε κάποια συμφωνία, κάποιο παζάρι. Λοιπόν, πέρα από τις μεταφορές και τον τουρισμό θα πρέπει να πείσετε την κοινή γνώμη και μπορείτε να το κάνετε αυτό με τον τρόπο που κάνει η Αμερικανική Γερουσία η οποία συνεδριάζει δημοσίως. Γιατί δεν το κάνει λοιπόν το Συμβούλιο Υπουργών. Ευχαριστώ κύριε Νιούτον Ντάν. Τώρα η κυρία Μπιλμπάου και μετά το Κρικέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τους εκπροσώπους της ε, Προεδρίας. Είχα μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλίας και δεν μπορούσα να ακούσω το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης. Έχω μια ερώτηση Μία, μία, μία μόνη ερωτησούλα. Όλοι συμφωνούμε με την Πράσινη Συμφωνία, την βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε παγίως τα προβλήματα των κρατών μελών ε, στο Συμβούλιο και ξεκινώ από τα TEN-T, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μιλάμε για κάποια έργα του 1994 δεν ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες εκείνες. Έχουμε επίσης αύξηση των εκπομπών από τα φερτηγά στις συνοριακές ζώνες. Επίσης έχουμε τις συνδυασμένες μεταφορές, έχουμε τις εναλλακτικέ ούτως ώστε να πετύχουμε τους ε, στόχους μας τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, το Γαλιλαίο, το τέταρτο πακέτο για σιδηροδρομικές μεταφορές που δεν ολοκληρώθηκε αυτό ούτε άρχισε να τρέχει όπως ε, είχαμε προσπαθήσει να γίνει στην προηγούμενη η ερώτηση είναι τι θα κάνετε στο Συμβούλιο, τι μπορείτε να κάνετε σε συνεργασία με το Συμβούλιο και με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε επιτέλους ε, τις προσπάθειές μας ε, και να πετύχουμε τους ε, σχετικούς δύο στόχους είναι λίγο φαρισαϊκό. Μιλάμε συνέχεια για πράσινη συμφωνία, μιλάμε για βιωσιμότητα, μιλάμε το πόσο μας και η βιωσιμότητα, η ψηφική τεχνολογία, αλλά έχουμε όλα αυτά τα σημαντικά προγράμματα και έργα τα οποία επίσης πάγια είναι σε παράλυση από πλευρά των κρατών μελών. Εσείς, Βλέπετε ότι το Συμβούλιο προτίθεται να κάνει κάποια βήματα προς εκείνη την κατεύθυνση. Εμείς συνεχώς προσπαθούμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Όχι, όχι, δεν, το λέω για να σας ε, επικρίνω εσάς προσωπικά. Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό, ε, ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί ο τουρισμός για το 2030, μπορούμε να φτάσουμε σε αύξηση μέχρι και 80%. Όμως, η Ευρώπη δεν είναι στέση να υποδεχθεί όλο αυτό τον κόσμο είναι θέμα βασικής υποδομής αυτό που αναφέρθηκε. Επίσης είπαμε για τη συνάντηση του Απριλίου και για κάποια πρωτοβουλία για βιώσιμο τουρισμό και θέλω να μου πείτε σε αυτή τη διάσκεψη που θα κάνετε τον Απρίλιο τι ρόλο έχουν οι περιφέρειες. Τα λέει συνέχεια η Επιτροπή των Περιφερειών. Θέλει να είναι παρούσα ε, για να γίνουν τα σχετικά. Και στην ε, χώρα των Βάσκων έχουμε πρόσφατη ανάπτυξη του τουρισμού και ακριβώς επειδή είναι φρέσκος ο τουρισμός χώρα των ε, ε, Βάσκων, έχει κάποια προβλήματα και ε, πρέπει να εμπλακούν όλοι οι συναρμόδιοι για να υπάρξει ε, πρόοδος και να υπάρξει και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε ένα σωρό επισκέπτες, χρειάζεται αμοιβαίο σεβασμός και αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει βιωσιμότητα, προσοχή στο κοινωνικό θέμα και στο περιβάλλον. Όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και όπως ξέρετε και εσείς όλα αυτά να πιάσουν τόπο σε επίπεδο περιφερειακό. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Ο κύριος Ντομινίκ Κρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους υπουργούς. Είπατε ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι τα δίκτυα. Η τροποποίηση το, των TNT και τα έξυπνα τεντή. Είμαι εισηγητή και για τις δύο εκθέσεις. Ε, συνεισηγητής με τον κύριο Μαρινέσκου ε, για το πρώτο θέμα και απλώς εισηγητή για το δεύτερο. Μόνος εισηγητή. Λοιπόν, είναι σημαντικό για να έχουμε πλήρη ενιαία αγορά για τα αγαθά και τους ανθρώπους, για να έχουμε την πράσινη ανάπτυξη και τον τις συνδυασμένε μεταφορές, να ρυθμίσουμε το θέμα το, της χρηματοδότησης. Αυτές οι εκθέσει λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικές και είναι και η προτεραιότητά σα. Η θέση του Συμβουλίου είναι μια μηδενική θέση. Νέο φαινόμενο. Δεν προτείνει τίποτα δηλαδή το Συμβούλιο. Όταν σας συνάντησα, μάλιστα, διερωτόμουν αν είχε νόημα να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο για μια θέση πάνω σε μια θέση όπως αυτή του Συμβουλίου, που είναι μηδενική. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή ένα τριμερή διάλογο με του συναδέλφου μέσα σε εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε συμφωνία, κατά τη γνώμη σα, πέστε μου. Οι θέσει είναι τόσο αποκλίνουσες που πραγματικά έχει νόημα να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Επίση, στην ε, Ευρώπη για να, δρομολογη... για να τελεσφορήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα χρειάζεται 8 χρόνια κατά όρο. Ε, και συχνά, επειδή υπάρχει τέτοιο περίπλοκες ε, διοικητικές διαδικασίες, δεν ξεκινάει ποτέ κανένα τέτοιο project. Ε, υπάρχει τεράστια απογοήτευση, γιατί η θέση του Συμβουλίου μου φαίνεται αδιανόητη. Δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε καθόλου. Δεύτερον, μιλήσατε πολύ για το, τις αερομεταφορές. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι δυστυχώς εκ μέρους του, ε, λόγω του Brexit, επειδή θα φύγει και το Γιβραλτάρ από το, τα προβλήματά μας, ας πούμε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μιλάμε για ένα ε, κείμενο, το σχετικό κείμενο, ε, το οποίο έχει μπλοκαριστεί εδώ και 7 χρόνια. Είναι τα σλότ, οι χρονοθυρίδες ε, των αεροπλάνων και πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο τραπέζι. τελευταίο θέμα τώρα, τουρισμός, Πρόεδρε. Πώς είναι δυνατόν Κάτι που όπως είπατε κι εσείς είναι περίπου το 10% του ΑΕΠ, 8% των, των θέσεων απασχόλησης και που υπάρχει στις συνθήκες όπως προνόμιο της Ευρώπης να μην έχει ούτε ένα ευρώ ως γραμμή προπολογισμού ανεξάρτητη. Αδιανόητο. Είναι λογικό να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, ας πούμε, και οι αερομετοφορέ που είναι συνδυάζονται με τον τουρισμό κτλ. Πώ είναι δυνατόν ο τουρισμός να μην έχει ούτε ένα ευρώ. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ε, καλεσμένους σας, ε, λέει η κυρία Τάλερ. Ε, ενδιαφέρονται αυτά τα οποία είπανε για το δίκτυο το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών πρόκειται για ένα πρόγραμμα 1,5-3 ε, εκατομμυρίου ευρώ και κάτι το οποίο αξίζει να αφήσουμε σκληρονομιά, αλλά δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι καταβάλλεται μεγάλες προσπαθίες για αυτό το θέμα για να ολοκληρωθεί το ζήτημα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ειδικά ως ε, μέλος ε, της Επιτροπής Βουλευτής από την Αυστρία. Θα χαρώ ιδιαίτερος γιατί αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα, ειδικά στη Δυτική Αυστρία. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξή: Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στο Συμβούλιο για το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και εάν ε, μπορούσατε να κάνετε μια ευχή, ποια ευχή θα κάνατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους και γείτονες ε, μόνο των Ούγγρων. Ήρθα επί τούτου στις Βρυξέλλες για αυτήν τη συνεδρίαση. Και το απόγευμα θα πρέπει να βρεθώ στην ε, Μαδρίτη σε μια άλλη συνάντηση. Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε το εξής. Ίσως οι βουλευτές, οι παρόντες εδώ, ίσως ε, δεν γνωρίζουν ότι κάθε έξι μήνες ε, όταν οι προεδρίες προετοιμάζουν την έντολή ε, τους, πάντα είναι αγώνας να περιληφθεί ο τουρισμός στο πρόγραμμα. Τώρα όμως η Κροατική Προεδρία εργάζεται εδώ και δύο χρόνια για να καταφέρει να ρίξει βάρος στον τουρισμό. Οι έξι μήνες αυτοί λοιπόν θα είναι μια πολύ σημαντική περίοδος και βεβαίω υπάρχουν οι συνάδελφοι που μπορούν να ενθαρρύνουν εδώ τους εκπροσώπους των κρατών μελών και θα δουν μια πολύ επιτυχημένη προεδρία νομίζω. Σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητέ Φράνο για τις προσπάθειές σας. Δύο συγκεκριμένα πράγματα τώρα ανα, τα αναφέρατε, αλλά δεν αρκεί να το αναφέρουμε. είναι η γραμμή στο ΠΔΠ για τον βιώσιμο τουρισμό. Εκεί πέρα θα χρειαστεί η στήριξή μας στην προατική κυβέρνηση, γιατί κάποιες άλλες κυβερνήσεις δεν θα το στηρίξουν. Θα χρειαστούμε λοιπόν την στήριξή σας εντός του Συμβουλίου και θα πρέπει να πείσουμε και την ε, Κομισιόν γιατί ακόμα δεν έχει ταχθεί με την πρόταση του Κοινοβουλίου. Ε, θα το διαπραγματευτούμε αυτό με τους υφυπουργού γιατί και στις συνοδοκορυφείς και στις άτυπες συναντήσεις θα έχουμε την ευκαιρία μετά αναφέρατε επίσης ε, τις ε, προσπάθειες ε, κοινού μάρκετινγκ προς τρίτες χώρες. Μπορείτε να μπείτε σε λεπτομέρειες γιατί κάποιοι συνάδελφοι βεβαίως θα βοηθηθούν από αυτήν την υπόθεση. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ κύριο Σφάιντερ τώρα. Και μετά η κυρία Κρούμπακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Έχω τρεις ερωτήσεις. Γιατί ήμουν ε, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου τώρα, είχαμε ψηφοφορία, οπότε ίσως επαναλάβω κάποιες ερωτήσεις ε, που έχουν ήδη γίνει. Πρώτα απ' όλα Ευρωβινιέτα. Ε, Δανία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία συμφώνησαν για μια κοινή βινιέτα, κοινό αυτοκόλλητο για την πληρωμή των διοδίων θα ήθελα λοιπόν άρα να σας ε, ρωτήσω εάν η Κροατία σκοπεύει κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας της ε, να ασχοληθεί και με τα ελαφρύτερα οχήματα, τα γιοταχή. Εγώ θα προτιμούσα να μην το κάνετε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι άποψη έχετε. Δεύτερον, για τους χορηγούς δεν έχουμε ακόμα μια πλήρη λίστα των χορηγών της Προεδρίας σας. Ε, εντάξει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να μας πείτε εάν κάποιοι από αυτούς τους χορηγούς σχετίζονται με την ε, Ευρωβινιέτα ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και το τρίτο ερώτημα, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών πάλι. Ε, υπάρχει πράγματι αυτή η μεγάλη προτεραιότητα τη σύνδεσης ε, των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών και ο περιορισμός κυκλοφορίας σε κάποιους ευρωπαϊκούς δρόμους. Εγώ προέρχομαι από την Άνω Αυστρία και Βεβαίω είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά εκεί στη μεθοριακή περιοχή. Δεν πειράζει αν δεν το ξέρετε συγκεκριμένα αλλά εντάξει μπορεί να μην μπορείτε να απαντήσετε απλά δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβετε τον συγκεκριμένο άξονα που είναι στην ε, Άνω Αυστρία εκεί. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρίνμπεργκ και μετά κυρία Ερμό. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, χαίρομαι ε, ιδιαίτερα που μας παρουσιάζεται το πρόγραμμα και έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Θα στηρίξετε το θέμα των δικαιωμάτων επιβατών ε, σιδηροδρόμων. Αφορά και τα δύο θέματα που αναφέρατε, δηλαδή την ε, διατροπικότητα, τη μετακίνηση των μεταφορών στο σιδηροδρόμους και τον βιώσιμο τουρισμό. Γιατί μόνο εάν ο κόσμος πραγματικά θεωρεί ότι τους παίρνουμε σοβαρά, δηλαδή αν δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τα δικαιώματα τους και στείλει αυτό το μήνυμα, ε, θα θεωρήσουν ότι τα εννοούμε αυτά τα οποία λέμε. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχουν τα ειστήρια. Στην περίπτωση που ε, δεν ταξιδεύουν ε, τα τρένα, αλλά και προσβασιμότητα για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, αλλά και για τα ποδήλατα που πρέπει να μπορούν να ανεβαίνουν στα τρένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να δείτε αυτό το θέμα αλλά και την ένταση που υπάρχει μεταξύ των ανέγγιχτων τοπίων ε, στον τουρισμό, αλλά και την βούληση επέκτασης του τουρισμού. Είναι μια αντίφαση. Ε, Παραδείγματο χάρη υπάρχουν ε, κάποια παραθαλασσία τοπία με πολύ μεγάλη δόμηση. Υπάρχουν βεβαίως άλλοι το οποίο που βλέπουμε ένα νέο δρόμο του βιώσιμου τουρισμού. Γιατί βεβαίως ε, λογικό είναι οι ντόπιοι να θελήσουν να επεκτείνουν τον τουρισμό όσο γίνεται, αλλά αν ε, δεν περιοριστεί αυτό δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτά τα τοπία. Σε ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. ακούσουμε τελευταία συνάδελφο. αυτή η νέα πράσινη συμφωνία είναι μια υπέρμετρη φιλοδοξία. Τη στιγμή που σήμερα δεν υλοποιούμε τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ήδη. Ε, να σας πω ποια προβλήματα έχουμε στην στο επίπεδο υποδομών των διευρωπαϊκών δικτύων. Στην Γερμανία και στη Σουηδία υπήρχαν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, τα οποία αποφασίστηκαν σε εθνικό επίπεδο για τις ιδεοτομικές μεταφορές και υποδομές. Και οι δύο χώρες ε, υποχρεώθηκαν να μειώσουν τις ε, πρικοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό, γιατί στη Γερμανία, ας πούμε, δεν έχουν αρκετούς μηχανικούς για να προχωρήσουμε αυτά που προβλέψανε. Έχουν ε, προβλέψει, μάλιστα, ε, να συνεργαστούν με Ρουμάνους μηχαν, μηχανικούς, ε, γιατί δεν έχουν αρκετούς ε, Γερμανούς. Στη Σουηδία αντίστοιχα προβλήματα, στη Γαλλία έχουν προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις. Όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα δεν προχωρούν. Στη Ρουμανία και στην Κροατία, όπως ξέρετε πολύ καλά την κατάσταση, τι προβλήματα υπάρχουν με το σιδηρόδρομο στην Ρουμανία. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τις αεροδομικές υποδομές και να απορροφήσουμε τα χρήματα. Την τελευταία περίοδο διάφορα δισεκατομμύρια δεν εκταμιεύθηκαν. Γιατί δεν ε, στηρίζει η Ευρώπη, δεν κάνει η Ευρώπη ό,τι κάνει οι Αμερικανοί. Κάνανε μια ομοσπονδιακή επιτροπή, ένα ε, ομοσπονδιακό φορέα, ας πούμε, για να επιτρέψει, να επιβλέψει όλη αυτή την προσπάθεια. Ε, εμείς, ας πούμε, εμείς ε, λέμε ότι όταν έχουμε τα χρήματα, α πούμε, τα πράγματα θα δρομολογηθούν από μόνα τους. Όχι, χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη στήριξη και πρόθεση. Όπως είπε και ο κύριος Ρικέ, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τα προβλήματα που υπάρχουν όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη για να προχωρήσουν τέτοια μεγάλα προγράμματα μαμούθ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ε, Επιτρέψατε μου και εμένα να κάνω μια ερώτηση. Είμαι σκιώδης ηγητής για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και ε, εδώ και χρόνια έχουμε κολλήσει. Δεν προχωράει τίποτα. Έχει κολλήσει το Συμβούλιο. Ε, εντάξει, η γη συνεχίζει να γυρίζει, αλλά έχουν κολλήσει οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μας. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρετε ως Κροατική Προεδρία να βρείτε έναν τρόπο για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση στο Συμβούλιο. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στηρίξετε και το Κοινοβουλίο. Έχουμε βρει μια θέση και είμαστε διατεθειμένοι να κινηθούμε με γρήγορες διαδικασίες για να επιτύχουμε πρόοδο, ειδικά στον Ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Γιατί είχαμε συζητήσεις για το πράσινο deal και τα λοιπά, το πόσο σημαντικό είναι να εξοικονομήσουμε διοξείδιο του άνθρακα. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα εδώ πέρα ε, που θα έπρεπε να μας απασχολεί πάρα πολύ. Μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η παράκλησή μου λοιπόν είναι η εξής. Ε, προωθήστε το. Φροντίστε να τοποθετηθεί εκ νέου η Κομισιόν και το Συμβούλιο για να πάμε από κοινού σε έναν τριμερή ε, διάλογο και να έχουμε αποτελέσματα σε ένα θέμα που έχουν συζητηθεί τα πάντα και πρέπει απλά να περάσουμε στην πράξη. Τώρα θα σας δώσω την δυνατότητα να απαντήσετε. Ο κύριος Μπίλεβερ, πρώτος. Ο κύριος Νομίζω ότι... Εγώ έχω τη μέρα του λέοντος από τις ερωτήσεις και όχι ο συνάδελφος προς τον τουρισμό, οπότε να σας πω για, το, για τις ε, μεταφορές και σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις που πραγματικά με χαροποιούν. Ε, εννοείται ότι θα πετύχουμε περισσότερα εάν συνεργαστούμε. Και για να δούμε τώρα να ομαδοποιήσουμε κάπω τι ε, ερωτήσει. Τάνια Σάτσου, το άρα που ακούσατε, Μπιτ, η Άσαν, η Κράτα, κουτό. Ε, Μία ομάδα απαντήσεων, ερωτήσεων συγγνώμη, τις καλύψαμε τώρα για να δούμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο και πιο σύντομα να σας τα πω τόσο ώστε και εσείς να έχετε το τοπίο ξεκάθαρο για το πώς θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και τα θέματα των επιβατών της αερομεταφορές σας απασχόλησαν και να προσπαθήσω να είμαι ε, ξεκάθαρος για τη γενική προσέγγιση που έχουμε για τους επιβάτες των αερομεταφορών είναι η εξή. Μια γενικευμένη, μια τέλο πάντων σφαιρική προσέγγιση κατά την ε, προεδρία μας. Δεν έχουμε πάρα πολλές προτεραιότητες. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτά που θεωρούμε ότι είναι πιο εφικτά και ένας από τους υλοποιείς στόχους είναι να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου όσον αφορά τις αερομεταφορές και να καλύψουμε και τα δικαιώματα των επιβατών Όσον αφορά δε τον ενιαίο ουρανό, ε, τώρα είναι στο χέρι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εμείς συνεχώς ε, συζητούμε με την Επιτροπή, διαπραγματευόμαστε και ε, σε κάνα μήνα θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα διατυπώσει καινούργια πρόταση, οπότε και θα αρχίσουμε τις επαφές σε επίπεδο κρατών μέλων και θέλουμε με Ουκρανία, Αρμενία και την Ισία να κλείσουμε κάποιες ε, συμφωνίες. Αυτά όλα στο εξάμεινο. Τώρα, όσον αφορά τα slots, και για αυτά γίνεται συζήτηση με την Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα τυπώσει μια οριστική πρόταση. Αυτά για τις αερομεταφορές. Τώρα, δεύτερη ομάδα ερωτήσεων για τους διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων και για τα ευφύ δίκτυα. Πρέπει να εμπλακούν όλα τα κράτη-μέλη, τα νέα κράτη-μέλη αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια για να είναι ανταγωνιστική η όλη ευρωπαϊκή οικονομία. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη ε, συνδεσιμότητα στις μεταφορές. Να διευρυνθεί επίσης το δίκτυο και έχουμε τάξει ως πρωτοβουλίες να ασχοληθούμε με τους υπάρχοντες διαδρόμους και επίσης να φροντίσουμε και για τα δίκτυα το Μάιο θα γίνει μια συνάντηση ε, κορυφής στη χώρα μας. Οπότε προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να έχουν και να κάποιες προτάσεις. Δεν είναι απλά τα πράγματα και το 2023 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή. Θέλουμε πάντως να έχουμε κάποια θεμέλια γερά για την υπόθεση αυτή, ούτως ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το δίκτυο και επίσης για τα δύο Ευρωπαϊκά δίκτυα θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα υπάρξει κάποια συμφωνία και επίσης ξέρουμε ότι έχει θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, αλλά υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και σε άλλα θέματα. Παρ' όλα αυτά κλείνονται συμφωνίες και για αυτό θεωρούμε ότι αν προσπαθήσουμε όλοι τελικά θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση πετυχημένη και ικανοποιητική. Ο κύριος Τελή με ερώτησε πώς θα υπάρξει σύνδεση με τα Δυτικά Βαλκάνια, γενικά τι συνδέσει θα γίνουν προς ε, νότιο-ανατολικά. Γι' αυτό και θέλουμε να υπάρχει ο διάδρομος της Αδριατικής, υπάρχει ε, μια πρωτοβουλία, ε, υπάρχει μια συμφωνία Αυστρίας, Σλοβανίας, Κροατίας και Σερβίας, ούτω ώστε να υπάρχει ένας νέος διάδρομος προς Δυτικά Βαλκάνια και έτσι θα έχουμε σύνδεση με την ε, Δυτική από τη μια και από την άλλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης, είχαμε ερωτήσεις για την Πράσινη Συμφωνία και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φτιάχνοντας νέο διάδρομο και προς Καρπάθια και αν αναπτύξουμε περισσότερο τον υπάρχοντα διάδρομο, αυτή η διάδρομη θα βοηθήσουν άπαξ και υπάρξει χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Καλύτερη συνδεσιμότητα θα έχουμε τότε. Θα έχουμε λιγότερες εκπομπές διοξιδίου. Επίσης, και η οικονομία θα αναπτυχθεί, θα γίνει πιο ανταγωνιστική στην διεθνή σκηνή. Επίσης θέλουμε να υπάρξει και ανάπτυξη των εμπορικών λιμένων, να υπάρχει σύνδεση των λιμένων ε, με σιδηρόδρομο, με εσωτερικές πλούτες οδούς, οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς τα εκεί. Έχουμε εμπειρία και ας είμαστε νέο κράτος μέλος. κύριε Φλέγκο, μας είπατε κάτι για την Αυστρία. την Ίστρια, την Ίστρια, συγγνώμη. Και υπάρχουν στατιστικά για το διοξίδιο. Τα έχουμε και στην Κροατία όπως υπάρχουν και αλλού και η χώρα ήδη έχει στραφεί στο πώς θα γίνουν επενδύσεις άνω του ενός δις. Έχουμε προετοιμαστεί για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και θέλουμε να υπάρχει αύξηση των επενδύσεων με πρόβλεψη άλλου ενός δισεκατομμυρίου. Φυσικά και θέλουμε ότι είναι πρόβλημα οι εκπομπές του διεξιδίου, αλλά επενδύουμε σε μορφές ε, μεταφορών που βοηθούν. Βοηθούμε επομένως την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά πρόσφατα μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη ε, και προβλήματα επίσης πρόσβασης στην χρηματοδότηση. Επίσης διασύνδεση νησιών, ε, βιωσιμότητα, ε, βέβαια θα ετοιμάσουμε την σχετική δήλωση και θα ζητήσουμε λιγότερο άνθρακα, περισσότερες επενδύσεις προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα, ιδίως όσον αφορά τη μόλυνση των θαλασσών από την ε, ναυσιπλοεία. Στη Βαλέτα το 17 συνήφθη μια συμφωνία και θέλουμε αυτή η συμφωνία να έχει συνέχεια. Επίσης, περιμένουμε νέες προτάσεις ε, επί τη βάση της Πράσινης Συμφωνίας και επίσης ρωτήσατε τι γίνεται με τις επενδύσεις στις υποδομές και πώς θα κάνουμε περισσότερα για τις ε, συνδρομικές μεταφορές σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία. Ε, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι κάθε επένδυση από τα ευρωπαϊκά ταμεία περνάει από πολλά φίλτρα και αυστηρό έλεγχο και δεν δίνεται έγκριση για επενδύσεις εάν υπάρχει επίπτωση αρνητική για το περιβάλλον. Γι' αυτό και γίνονται σχετικές μελέτες. Γνωρίζουμε ότι το έργο αυτό είναι δύσκολο, αλλά οπωσδήποτε συμφωνούμε ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες. Όσο αφορά τα δικαιώματα των επιβατών τώρα, στους σιδηροδρόμους. Επαναλαμβάνω, η γενικότερη προσέγγιση εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο. Και τώρα περάσαμε στη φάση των συζητήσεων. Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα θα υπάρξει μια συμβαστική λύση, τόσο ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες του Συμβουλίου, θα σας πω πολύ σύντομα το εξή. Ο τρόπος που εργάζεται το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτή την ευθύνη δεν τη φέρει μόνο το κράτος προεδρία αλλά όλα τα κράτη-μέλη. Και η Κομισιόν εξάλλου. Αλλά και οι ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι η βασική δραστηριότητα ασκείται εδώ μέσα, αλλά πρέπει να υπάρχει και δράση στα κράτη-μέλη μας. Γιατί μόνο αν δράσουμε από κοινού θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε, ούτω ώστε να υπάρχει και διαφάνεια της εργασίας και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και να υπάρξει και πλησίασμα ε, των θεσμικών οργάνων ε, προς τον πολίτη όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή της Προεδρίας μας προσπαθούμε να δείξουμε ανοιχτό πρόσωπο ε, προς το κοινό, στα ΜΜΕ και στην Κροατία. Οργανώσαμε διάφορες συνεντεύξεις τύπου για να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες μας και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεχάσουμε να λογοδοτήσουμε για την πρόοδο που θα σημειώσουμε για όλα τα θέματα και τα οποία συζητάμε. Είναι υποχρέωσή μας αυτή απέναντι στους πολίτες μας. Ακούστηκαν πολλοί άριθμες ερωτήσεις, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να κατάφερα να σας απαντήσω αρκετά συγκεκριμένα. Αν κάποιος παρόλα αυτά επιθυμεί να συνεχίσει τις ερωτήσεις, μπορούμε να συνεχίσουμε και κατηδίαν, κατά μόνας. Και ο επόμενος ε, υπουργός, ελπίζω να είμαι λίγο πιο σύντομος από τον ε, ομολογό μου τον κύριο Μπιλαβέρ, θα απαντήσω ομαδικά σε διάφορες ερωτήσεις, γιατί διάφοροι βουλευτές επανέλαβαν κάποια θέματα. Πάντως, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους σας για την πρωτοβουλία να υπάρξει μια νέα γραμμή προϋπολογισμού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο δεν υπάρχει έγκριση για κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα για να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο. Εξού και η σημασία σας, η σημασία της δράσης σας για να προτάξουμε τον τουρισμό. Εμείς Θέλουμε να δώσουμε καλύτερη θέση στον τουρισμό. Ο κύριος Μπιλαβέρ μίλησε για αυτό το θέμα. Εγώ θα το αγγίξω πολύ σύντομα. Καταρχάς έχουμε την Σύνοδο Κορυφή στο Ζάγκρεπ του Μαΐου για τη διεύρυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ανοιχτή αυτή η προοπτική για όλα τα κράτη-μέλη που δεν είναι, για τα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, ε, μαύρες τρύπες Εντό της Ευρώπης ε, ή στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι α πούμε τα Δυτικά Βαλκάνια αυτή τη στιγμή, μια μαύρη τρύπα. Ε, τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων επιθυμούν να γίνουν μέλη. Και ελπίζω οι διαπραγματεύσει με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία να ξεκινήσουν γρήγορα και η Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ να επιβεβαιώσει αυτή την προοπτική. Επίση, πολλέ από τι ερωτήσει αφορούσαν τι μεταφορέ και άλλα θέματα. Νομίζω ότι αυτά θα μπορούσαν να συζητηθούν ε, και να επιληθούν στις διαπραγματεύσεις αυτές, στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου, για να χρηματοδοτήσουμε και να στηρίξουμε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα Ενιαία Αγορά, Single Market, όλοι οι μηχανισμοί δεν είναι ακόμη στη διάθεσή μας, ούτε έχουν εξαντληθεί. Θέλω την ε, υποστήριξή σας. Ο κύριος Φλέγκο και ο κύριος Ίστβαντ, που είναι φίλος και θα βρεθούμε στη Μαδρίτη ως Υπουργοί Τουρισμού και θα ενημερωθούμε για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ίστβαν, που αναγνωρίζεις την ανάγκη αυτή να θέσουμε τον τουρισμό στο κέντρο των ανησυχιών μας νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε ό,τι αφορά τις, τα κοινά δρομολόγια που έθιξαν και ο κ. Ίστβαν και ο κ. Φλεγκό, για να υπάρχει ε, καλύτερη διασύνδεση με τις μακρινές αγορές. Υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη που έχουν εμπειρία σχετική και που έχουν ε, παρόμοιες προσεγγίσεις. το χάρη με την κινέζικη ή με την κορεατική αγορά. Υπάρχει μια πρακτική ομαδικών ταξιδίων ούτω ώστε να μπορέσουμε να επισκεφθούμε πολλά κράτη στην ίδια επίσκεψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη δράση, ούτω ώστε να παρουσιάσουμε την Ευρώπη πιο αποτελεσματικά σε αυτέ τι μακρινέ αγορέ. Επίση μιλήσαμε για την, ε, το σημαντικό δυναμικό του τουρισμού και το δυναμικό ανάπτυξη. Η κυρία Οτεγό το ανέφερε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι το 2030 η ανάπτυξη του τουρισμού θα είναι πολύ σημαντική. Όλη η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να συμμετάσχει ε, σε αυτή την ανάπτυξη. Υπάρχουν διάφοροι προορισμοί, φυσικά, και κάθε χώρα, ας πούμε, προβάλλει με το δικό της τρόπο τον τουρισμό. Το θέμα είναι να υπάρχει μια διαφοροποιημένη ζήτηση τουριστικού τύπου. Θα πρέπει δηλαδή να κατευθύνουμε κάποιες τουριστικές ροές προς νέους προορισμούς, προς την Ήπεθρο περιφήν ε, και για να ελαφρύνουμε τους προορισμούς που δέχονται πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά και έχουν μείνει πίσω τουριστικά. Να τις βοηθήσουμε δηλαδή. Να γίνει αυτή η διαφοροποίηση ε, και να πούμε σε αυτούς που έρχονται και μας ε, επισκέπτονται ποιοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν ατελείωτο κόσμο και ποιοι είναι σχεδόν άδειοι και καλό θα ήταν ας πούμε ενδεχομένως να του επιλέξουν για να τις ανακαλύψουν αυτές τις περιοχές, ε, για να ανακαλύψουν νέους προορισμούς. Επίσης, μιλήσαμε για τη διαφάνεια στις αποφάσεις του Συμβουλίου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει το Συμβούλιο, προφανώς. Και νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία σας για μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις του Συμβουλίου. Όπως ακριβώς στο Κοινοβούλιο που υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Και όχι μόνο στις ψηφοφορίες, αλλά στις συζητήσεις γενικά. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η προσπάθεια να εξασφαλίσω μεγαλύτερη διαφάνεια στις εργασίες του Συμβουλίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολο να δούμε Πού υπάρχουν αμφιβολίες, πού υπάρχουν ε, σκιές, πού υπάρχουν παρεξηγήσεις ναι. με κάποια κρατημέλη και με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό πιο αποτελεσματικά, ε, αν χρειαστεί και με διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τους Εθνικούς Βουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα και σίγουρα θα δώσει σημασία το Συμβούλιο σε αυτή την πρωτοβουλία σας. Σε ό,τι αφορά τον σιδηροδρομικό κλάδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, μιλήσατε πάρα πολύ ε, για την ποιοτική ε, διάσταση του κλάδου αυτού. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το να δημιουργήσουμε νέους διαδρομικούς άξονες τόσο, όσο να βελτιώσουμε την ποιότητα και την, να, αυξήσουμε την ταχύτητα στα κομμάτια που έχουμε ήδη σειροδρομική κάλυψη. Ο κύριος Πτεγκό ε, έθιξε αυτό το θέμα πολύ εύγλωτα. Ε, μερικές φορές για 300 χιλιόμετρα χρειαζόμαστε 5, 10, 12 ώρες. Ειδικά στην Δυτική Ευρώπη το να φτάσουμε σε ταχύτητες 300 χιλιόμετρων είναι αδιανόητο ας πούμε. Ε, όταν φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε ας πούμε ποδήλατο με σιδηρόδρομο Φερρυπίν και χάρη στο σιδηρόδρομο να πλησιάσουμε σε πολλές ε, και διάφορες περιοχές. Αυτό ο συνδυασμό των ποδηλατοδρόμων με τους σιδηροδρόμου είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό του σιδηροδρομικού τομέα. Γιατί συνδέεται και με την ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό το κομμάτι. Ο σιδηρόδρομος δηλαδή. Επίσης, η φυσική μας πόρη και πλούτος είναι η αιτία που είμαστε τουριστικός προορισμός. Θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε και τις φυσικές και τις πολιτιστικές ε, ομορφιές. Από αυτό εξαρτάται η ανάπτυξη του τουρισμού μας. Θα πρέπει λοιπόν να, έχει, να τις πλησιάσουμε με βιώσιμο τρόπο για να έχουμε και βιώσιμο τουρισμό. Για να προστατεύσουμε το, τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Και άρα μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να είναι βιώσιμη για να δημιουργηθούν νέες δουλειές. και για να μπορέσει ο κόσμος να ζει κανονική ζωή στις ε, τουριστικές περιοχές και οπωσδήποτε χρειάζονται μέσα μεταφοράς ε, που θα βοηθούν τους τουρίστες ε, να φτάνουν στους προορισμούς με τρόπο σύγχρονο, πολιτισμένο και βιώσιμο. Ελπίζω λοιπόν η συζήτηση αυτή να συνεισφέρει στα συμπεράσματά μας τον Μάιο και όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών τον ε, Μάρτιο θα γίνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην βιωσιμότητα του τουρισμού, παρουσία τοπικών εκπροσώπων που θα συζητήσουν την περιοχή του Δούναβη που θα είναι το βασικό θέμα και την ανάπτυξη του τουρισμού σε διάφορες άλλες περιοχές της Υπέθρου. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω και η στήριξή σας ε, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς και για τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες. Και αύριο στη Μαδρίτη θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τρόπο ουσιαστικό έτσι ώστε ο τουρισμός να γίνει πιο βιώσιμος καθώς επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάτουσιτς και κύριε Μπίλεβερ. Όπως βλέπετε η Επιτροπή μας γνωρίζει τα θέματα, έχει εμπειρία και είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στην επιτυχία της Κροατικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εκμεταλλευτείτε αυτήν τη γνώση και την εμπειρία γιατί τελικά η δική σας η επιτυχία είναι και δική μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτήν την επικοδομητική συζήτηση σήμερα. Θα συνεχίσουμε στις 2.30. Θα συνομιλήσουμε με τους Ευρωπαίους συντονιστές των διευρωπαϊκών δικτύων. Η κυρία Ανταλή θα με αντικαταστήσει από το απόγευμα και μετά. Γεια σας.